Έχουμε πέντε μέλη. Απαρτία μπορούμε να ξεκινήσουμε. Share with you first is the... Λοιπόν, να σας πω τα αποτελέσματα των αποφάσεων των συντονιστών. Θα μπορούσε να είναι απόλυτα νιαρό αυτό, αλλά δυστυχώς είμαι υποχρεωμένη να σας τα διαβάσω έτσι, για τα πρακτικά. Προσοχή λοιπόν. Σήμερα το πρωί λάβαμε αποφάσεις για αιτήματα για ε, ημερήσεις διατάξει των επόμενων συνεδριάσεων, ε, ε, τις αναφορές ε, για την Αφρική. Ε, επίσης, ε, αναφορές ε, για το, την υπερταχεία στην Ισπανία θα προσθεθούν στην ημερήσια διάταξη και επίσης ε, ε, συμφωνήθηκαν και κάποια ακόμα θέματα για εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις. Αποφασίσαμε να υποβάλουμε γνωμοδότηση στη νέα ε, νομοθετική έκθεση της ΑΦΚΟ για την πρόταση για την πρωτοβουλία των πολιτών, την νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ζητήσουμε και την χρήση του άρθρου 54. Τώρα, Κάποιες συστάσεις έκλεισαν ε, κατόπιν προτάσεώς μου, ε, η 0397, η 0400, η 0401 θα κλείσει, 0431 και η 0499 θα ε, θεωρηθεί παραδεκτή και θα κλείσει αμέσως. Τώρα, διερευνητικές επισκέψεις θα γίνει μία στο πρώτο εξάμεινο του 2018 το Φεβρουάριο, στη διάρκεια της τυρκουάς εβδομάδας, στην ε, περιοχή Βάουτσεν της Γερμανίας ε, και υπάρχει και η πιθανότητα να διοργανωθεί μια ακόμα συνεδρίαση σε περίπτωση που λάβουμε εξαίρεση για να μπορέσουμε να οργανώσουμε ε, αποστολή εκτός ε, ε, πράσινης εβδομάδας. Σε αυτή την περίπτωση η αποστολή θα γίνει Πέμπτη Παρασκευή. Για τις ε, δημόσιες ακροάσεις αποφασίσαμε να γίνει μία για τους ενδοκρινικές διαταράκτες και τις επιπτώσεις του στην υγεία και το περιβάλλον που θα γίνει την άνοιξη του 2018 και θα προσκαλέσουμε και την Επιτροπή ΕΜΒΗ για να συμμετέχει και αυτή στην ακρόαση. Υπάρχει και μία ακόμα, ε, η επισφαλής εργασία, η οποία θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου και ε, θα εγκρίναμε και το επικαιροποιημένο σχέδιο προγράμματος και ζητήσαμε από τη Γραμματεία να ε, δει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες όσον αφορά την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου. Αποφασίστηκε η Γραμματεία να καταρτήσει ένα σχέδιο κειμένου για το ε, δημοσίευση του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάποια βασικά θέματα. Ενημερώσαμε επίσης τους συντονιστές για την ε, συνεδρίαση ε, Petty Network και τη συνεδρίαση Cluster με το Σώμα των Επιτρόπων, επί ενημέρωσα για όλα αυτά και αποφασίσαμε ε, κάποια περαιτέρω θέματα για ε, παραγγελία μελέτης για το φορολογική συμμάρφωση το λεγόμενο φάτικα και επίσης κάποια θέματα αναβλήθηκαν για την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Αυτά λοιπόν. Τώρα, για την διερευνητική επίσκεψη στη Μαδρίτη, στην Ισπανία, που έγινε το Μάιο ε, φέτος, η κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας και θα της δώσω αμέσως το λόγο για να σας ενημερώσει για το θέμα αυτό. Έχουμε εδώ μαζί μας ε, και εκπροσώπους από την Ισπανία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Τζούτ λοιπόν έχει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Σεσίλια. Την αρχική έκθεση την έκανα στις 30 Μαΐου στην Επιτροπή, λίγες μέρες μετά την επιστροφή μας από τη Μαδρίτη και τα πάντα ήταν πολύ νοπά. Ε, ήταν πολύ έντονο αυτό το διήμερο το οποίο περάσαμε στην ε, Ισπανία. Εξετάσαμε διάφορες ε, ιστορικές υποθέσεις για απαγωγή νεογέννητων από νοσοκομεία και από κέντρα και με ευτήρια στην Ισπανία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και υπήρχαν και πολλές αναφορές για το θέμα αυτό. Στην ε, έκθεση αυτή τότε ε, τόνισα πόσο συναισθηματικά φορτισμένη και έντονη ήταν αυτή η επίσκεψη. Αυτό το σκάνδαλο των απογωγών παιδιών ε, στη διάρκεια της δικτατορίας αλλά και μετά με τη μετάβαση στο Δημοκρατία αναγνωρίστηκε από όλους εκείνους που συναντήσαμε. Υπήρχαν βέβαια κάποιες διαφορές μεταξύ θυμάτων, αρχών, δικηγόρων και ε, οι διαφορές αφορούσαν τον αριθμό των ατόμων που ε, τους επηρέασε αυτό το σκάνδαλο, αν πρόκειται για οργανωμένο δίκτυο ή αν ήταν μεμονωμένα άτομα, αν έγιναν αρκετά προκειμένου να υποστηρίξουμε τις έρευνες ε, για τις φερόμενες απογωγές παιδιών και για τη στήριξη των θυμάτων, είτε πρόκειται για νομική στήριξη ή για ψυχολογική στήριξη των ατόμων που επλήγησαν. Ε, από τότε, ε, από το τέλος Μαΐου και μετά, συνεργαζόμαστε με τη Γραμματεία και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Καρολίνα στην Γραμματεία της Επιτροπής. Ε, εργαστήκαμε σκληρά για να καταρτήσουμε ένα σχέδιο έκθεσης, το οποίο θα έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων όσων συμμετείχαν στην διερευνητική αποστολή. Και ο στόχος είναι να ε, δούμε τα πράγματα και να τα καταγράψουμε κατά λέξη. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε τα περισσότερα ε, γιατί ξέρουμε ότι θέλουν ε, όλοι να έχουν τις λεπτομέρειες και μετά από τη συζήτηση με τις αρχές και θέλουμε λοιπόν να αναφέρουμε όλες τις συναντήσεις που είχαμε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την Ισπανική Εκκλησία, με τον Ισπανό Δημοσιολαβητή, την ε, Αρμόδια Επιτροπή στο Ισπανικό Κοινοβούλιο, με τους αναφέροντες, ε, με ομάδες θυμάτων, ε, δημοσιογράφους που κάνουν έρευνα και νομικούς που συμμετέχουν στην όλη διαδικασία για να διαπιστώσουν τι συνέβη σε αυτές τις περιπτώσεις. Προσπαθήσαμε και νομίζω ότι υπήρχε και πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της Επιτροπής και τους ευχαριστώ ε, και με τη συμφωνία όλων ε, καταρτίστηκε αυτή η έκθεση για την ε, αποστολή και έχουμε καταλήξει σε 15 συστάσεις οι οποίες πρέπει να συζητηθούν από την Επιτροπή, να τροποποιηθούν και να τις συμφωνήσουμε στη συνέχεια. Πριν ξεκινήσει η συζήτηση για αυτές τις συστάσεις, ε, στις οποίες ε, γίνονται πολύ συγκεκριμένες ε, συστάσεις προς την Ισπανική κυβέρνηση για δυνατότητες για τεστ DNA, καλύτερη στήριξη προς τα θύματα, μια ιδιωτική ερευνητική επιτροπή που θα εξετάσει τι συνέβη σε αυτές τις υποθέσεις, συγκεκριμένες συστάσεις προς την Ισπανική Εκκλησία για να ανοίξουν τα μητρώα τους και να τα διαθέσουν ε, ε, για τα θύματα τα οποία ερευνούν και αναζητούν τα μέλη της οικογένειάς τους και το τι απέγιναν. Και πριν ε, ξεκινήσει η συζήτηση για αυτές τις συστάσεις, θα ήθελα να ολοκληρώσω ε, αποτείοντας φορό τιμής ε, στους αναφέροντες που ήρθαν εδώ στην Επιτροπή, διότι διαδραμάτισαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και για τη διεξαγωγή αυτής της αποστολής. Ε, συναντήσαμε αρκετά θύματα όταν ήμασταν εκεί στη Μαδρίτη και νομίζω ότι πρέπει ε, να αναφέρουμε τον πόνο και τα χρόνια που έκαναν σε αυτοί οι άνθρωποι ε, πολλοί εξ αυτών ε, ε, σπατάλησαν χρόνια ζητώντας στοιχειώδη πράγματα. Τι απέγινε με τους ανθρώπους που έχασαν, είτε ήταν παιδιά, αδέρφια ή και γονείς όταν κάποιος διαπιστώνει ότι είναι υιοθετημένο με τέτοιο τρόπο ε, απατηλό. Και αυτές τις ιστορίες πρέπει να τις έχουμε κατά νου όταν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτές τις εργασίες και πρέπει να βρίσκονται στο μυαλό μας ε, κάθε φορά που θα προχωρούμε και θα ζητούμε μια ισχυρή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι πολύ συχνά διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ε, πραγματικά βίωσαν πολύ προσωπικό πόνο. Μία γυναίκα μας είπε ότι ένιωσε ότι θα πεθάνει από τη ραγισμένη της καρδιά και όχι από τα γεράματα λόγω του πόνου που ένιωσε. Ε, και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να ακούγονται ε, ε, προφανή, αλλά αυτή είναι η ζωή πραγματικών ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά βίωσαν πόνο και υπέφεραν και όπου μπορούμε να τους βοηθήσουμε να λάβουν απαντήσεις, πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να τους βοηθήσουμε. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε αυτή την έκθεση για να έχουμε απτά αποτελέσματα και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε από εκεί και πέρα το διάλογο και με τις δημόσιες αρχές και με τις ε, αρχές της Εκκλησίας στην Ισπανία. Ευχαριστώ και να τονίσω και εγώ ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τη Γραμματεία και κυρίως τη Καρολίνα που έκανε εξαιρετική δουλειά για το θέμα αυτό. Και επίση θα ήθελα και εγώ εξ ονόματο της Επιτροπής να σε ευχαριστήσω Τζουτ γιατί ήσουν επικεφαλής αυτή τη πάρα πολύ ευαίσθητη διερευνητική αποστολή και ε, έγινε αυτό με την υποστήριξη συναδέλφων και με την ε, ευαισθησία που χρειάζεται. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και για το σεβασμό που επέδειξες προς όλους εκείνους που ε, ε, νεπλάξαν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος τώρα το λόγο για το θέμα αυτό. Είναι εδώ οι σκιώδεις ε, εισηγητές, η κυρία Πιτέρα. Ευχαριστώ πολύ. Συμμερίζομαι τη θέση σας, κύριε Πρόεδρε, ότι ήταν πολύ δύσκολη αυτή η επίσκεψη και λάβαμε πολλές ε, ε, αμφίσμες πληροφορίες. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν ε, θα πρέπει να έχουμε αφελείς και πολύ και πολύ μονόπλευρες ε, θέσεις. Ε, είναι πολύ δύσκολο το θέμα, διότι κάποια άτομα ή ακόμα και κλιματικές οργανώσεις ε, μπορεί να, να ενήργησαν, μπορεί να υπάρχουν και κάποια οικονομικά ωφέλη, να έχουν χτιστεί νοσοκομεία λόγω αυτών των υιοθεσιών. Θα πρέπει να φροντίσουμε να διατηρήσουμε ισορροπημένη προσέγγιση στο θέμα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες που μας επιτρέπουν να περιγράψουμε την κατάσταση και γνωρίζουμε ότι εφόσον οι ισπανικές αρχές δεν διαλευκάνουν το θέμα. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε τι πρέπει να γίνει. Χρειαζόμαστε όλα τα γεγονότα ε, προτού να μπορούμε να πάρουμε θέση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να ζητάει κανεί το λόγο από όσου ήταν στην αποστολή. Α, ναι, η Ελεονόρα, παρακαλώ. Ε, Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Να τονίσω και εγώ την εξαιρετική συνεργασία για μια πρόταση τελικά η οποία θα έλεγα σέβεται ε, την πραγματικότητα αυτής της αποστολής. Νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε κάπως τα θέματα αυτά. Και εγώ σημείωσα τεράστια κενά και τεράστιες αντιφάσεις ανάμεσα στις αρχές τις οποίες συναντήσαμε. Για μας ε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σύμπτωμα, αν θέλετε, μιας κατάστασης η οποία δεν μπορεί παρά να ληφθεί υπόψη. Στην ουσία διαπιστώσαμε ότι οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στις ισπανικές αρχές, οι οποίες δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν όπως θα έπρεπε τις έρευνες και δεν είναι σε θέση προληπτικά θα έλεγα να πάρουν τα μέτρα τα οποία απαιτούνται. Καταρχάς θα πρέπει να αναφερθούμε στις υποχρεώσεις τις οποίες έχει σε επίπεδο διεθνού συνταγματικού δικαίου η Ισπανία όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των ανηλίκων και φυσικά οι συμβάσεις για την προστασία από ε, απαγωγές και τα Έχουμε λοιπόν την υπόθεση που ονομάζουμε συνολικά η περίοδος Stolen Babies ήταν κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό σαν φαινόμενο κατά τη διάρκεια της περίοδου του Φράνκο και νομίζω ότι τα εγκλήματα αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν και συλλογικού τύπου γιατί είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλαπλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουμε να κάνουμε με μια οργάνωση η οποία παρενέβη για να οργανώσει τις απαγωγές αυτές. Η Ισπανία θα πρέπει, θα πρέπει έλεγα, να <clears throat> επικυρώσει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και έτσι θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν ακριβώς τέτοιου είδους εγκλήματα ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εμείς ε, ζητήσαμε από τις ε, Ισπανικές αρχές να μας πούν ποια είναι σήμερα η κατάσταση των ε, συστάσεων του ΟΗΕ που είχαν προταθεί στις Ισπανικές αρχές το 2014. Σε αυτό το αίτημα δεν πήραμε ποτέ καμία απάντηση. Και τέλος η περίπτωση των παιδιών που έπεσαν θύματα απαγωγής κατά τη διάρκεια της περίοδου του Φράνκο ε, θα πρέπει ε, στα πλαίσια να υπάρξουν διορθώσεις στα πλαίσια του Ισπανικού νόμου για την αμνηστία ε, ένα νόμο τον οποίο ο ΙΕ το 14 ζήτησε να καταργηθεί και να αντικατασταθεί και θα έλεγα υπάρχουν και μία σειρά άλλων θεμάτων τα οποία στην παρούσα φάση τουλάχιστον δεν είμαστε σε θέση να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, ξέρω ότι αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο όλοι θα ήθελαν να πούνε πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα ήθελα παρακαλώ να ακούμε τι λέει ο ένας στον άλλον και να μην επαναλαμβάνουμε αυτά τα οποία έχουν ήδη υποθεί. Η κυρία Σντάνοκα έχει το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομη. Να ευχαριστήσω την πρόεδρο της αποστολής μας. Ήδη ανέφερε τα βασικά θέματα και συμφωνούμε απολύτως με το επεξηγηματικό τμήμα της έκθεσης θα υποβάλουμε ε, τροπολογίες ε, όσον αφορά τις συστάσεις. Νομίζω ότι η βασική ε, το βασικό ζήτημα για το οποίο υπάρχουν διαφωνίες είναι το αν ήταν τυχαία ή συστηματική ε, αυτή η πρακτική. Εγώ νομίζω ότι ήταν ε, συστηματική και θα πρέπει να την κρίνουμε ως τέτοια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλπιόλ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο λοιπόν της αντιπροσωπείας για όλη την προσπάθεια την οποία έκανε έτσι ώστε να υπάρξει μια κάποια συνένεση και ήθελα να την ευχαριστήσω και για τον δραστήριο ρόλο της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά επίσης για την επικοινωνία που είχε με τους αναφέροντες όπως επίσης και με τις ενώσεις των θυμάτων του συλλόγου των θυμάτων <clears throat> έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Έχω την εντύπωση ότι η αποστολή αυτή οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα. Εμείς καταφέραμε να θέσουμε σε επίπεδο πολιτικής συζήτηση το θέμα των απαγωγών των παιδιών. Χάρη σε αυτές τις αναφορές πρέπει να το απογραμμίσουμε. Και είναι επίσης σημαντικό ότι η έκθεση υπογραμμίζει επίσης γιατί ήρθαν οι αναφέροντες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί ένιωσαν την εγκατάλειψη, την ανικανότητα και την αδράνεια των αρμόδιων Ισπανικών αρχών και της Ισπανικής Εκκλησίας. Υπήρξε έλλειψη έρευνα στην Ισπανία, δεν υπήρξε ανταπόκριση στα αιτήματά τους και γι' αυτό οδηγήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εφόσον λοιπόν ίσχυσαν αυτά τα οποία είπαμε αναγκάστηκαν να έρθουν στις Βρυξέλλες. Πρέπει να πούμε εμείς ότι το Ισπανικό κράτος δεν ασχολήθηκε και δεν χαρακτήρισε εκ των υστέρων τις υποθέσεις αυτές ως βίαιες απαγωγές. Ε, το θέμα αυτό έχει συζητηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου και στην ομάδα των Ηνωμένων Εθνών ειδικά για τα θέματα ε, των θυμάτων ε, απαγωγών, βίων απαγωγών. είναι κάτι το οποίο κάνει αυτή την προσπάθεια, ζητά μάλλον να γίνει η προσπάθεια που πρέπει και από τις Ισπανικές αρχές. Εμείς κατά τη διάρκεια της τροπολόγησης του κειμένου θα καταφέσουμε κάποιες προτάσεις. Υπάρχει εδώ η ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε ότι υπήρχε ένα συστηματικό πρόγραμμα με συγκεκριμένες ευθύνες, με ευθύνες επίσης και των δημοσίων αρχών. Και αυτό ακριβώς εξηγεί το γιατί υπήρξαν κλοπές, κλοπές, απαγωγές παιδιών για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα θέσουμε και άλλα θέματα μέσω τροπολογιών, σαν παράδειγμα οι αποδείξεις μέσω της μεθόδου ADN να είναι αποδείξεις δωρεάν για όλους τους εμπλεκομένους. Να διευκρινιστεί ο ρόλος και να διασφαλιστεί η συνεργασία της Εκκλησίας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 ευχαριστήσω και εγώ να πω ότι συμφωνώ γενικά με τις προτάσεις. Ελπίζω ότι οι τροπολογίες που θα κατατεθούν θα σέβονται την βασική γραμμή την οποία ακολουθείς στην έκθεσή σου. Πιστεύω ότι είναι μια έκθεση εξισορροπημένη Ελπίζω να μην υπάρξει υπερβολική πολιτικοποίηση μέσω των τροπολογιών της υπόθεσης αυτής, να έχουμε στο τέλος ε, μια έκθεση, όπως είπε η κυρία Αλμπόλ, να μην προσπαθήσουμε να επιτεθούμε πολιτικά σε διάφορες ομάδες, η εκκλησία κτλ. Νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια και συμφωνούμε με τη γραμμή πάντως την οποία ακολούθησε η Πρόεδρος. Τώρα για το αν είναι οργανωμένη η προσπάθεια αυτή για τις απαγωγές και τα λοιπά. Νομίζω ότι οι ισπανικές εισαγγελίε έχουν ανακρίνει τα θέματα αυτά σε πολλαπλές φάσεις και με διάφορους εμπλεκομένους για τα τελευταία 40 χρόνια. Υπάρχουν αμφιβολίες λοιπόν για το αν πράγματι ε, είναι κάτι το οργανωμένο. Εγώ δεν θα αντικαταστήσω εδώ τους ε, ανακριτές και τους δικαστές. Εγώ πιστεύω στην ε, ανεξαρτησία της ισπανικής δικαιοσύνης που λειτουργεί μέσα σε μια δημοκρατική χώρα. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ε, αυτά τα οποία ισχυρίστηκε η κυρία Αλμπιόλ. Νομίζω ότι πάρα πολλές δημόσιες αρχές και υπηρεσίες στην Ισπανία είναι ανεξάρτητες και εν πάση περιπτώσει εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Χαίρομαι που όλοι όσοι συμμετείχαν λίγο πολύ μπορούν να συμφωνήσουν με αυτά που περιέγραψε η επικεφαλής της αποστολής. Κάτι που ε, διευκολύνει τόσο τη δουλειά μας εδώ. Ε, δείχνουμε αξιοπρεπές πρόσωπο απέναντι στους αναφέροντες που είναι και παρόντες. Θα πρέπει πάντα να επιδεικνύουμε σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που έχουν υποφέρει τόσο. Έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάργαρετ Τουίτ. Μπορεί να μην πρόφερα σωστά το όνομά σας. Πείτε μου πώς προφέρετε σωστά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τσιούτ λέμε στην Ιρλανδία, όπως τη λέξη Institute. Αλλά ναι, έχουν ακούσει πολλά τα αυτιά μου. Σας ευχαριστώ για αυτήν την ε, ε, ενδιαφέρουσα και αναλυτική έκθεση. Γίνονται πολλές αναφορές στην υποστήριξη προς τα θύματα και τα δικαιώματα των ε, θυμάτων. Συνομίλησα ε, με ε, τον συνάδελφο αρμόδιο για την οδηγία 2012-29 που είναι η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων. Τελευταία φορά που συνομιλήσαμε σε τούτη την αίθουσα ήταν ε, το 2015 και η οδηγία αυτή τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2015. Μπορεί λοιπόν να ισχύει η οδηγία στην περίπτωση αυτή εφόσον η ποινική διαδικασία πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία μεταφοράς ε, στο ε, Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας που ήταν η 15η Νοεμβρίου. Ακόμα και και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί τα εγκλήματα αυτά πριν πολλά χρόνια, τα θύματα δικαιούνται προστασία σύμφωνα με την ε, οδηγία αυτή. Αυτό σημαίνει ότι ισχύει για οποιαδήποτε ποινική διαδικασία έχει ξεκινήσει. Υπάρχουν υποθέσεις που ανοίξαν το 2016, τρεις υποθέσεις το 2017 και ε, αναφέρονται στη σελίδα 13 και πολλές ε, υποθέσεις που εκκρεμούν ακόμα. Η οδηγία λοιπόν ισχύει για όλες αυτές ε, τις υποθέσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι να αναφερθούμε σε υποθέσεις ε, πριν ε, το, που είχαν κλείσει πριν τις 15 ε, Νοεμβρίου του 2015. Πρόεδρος, ε, σας ευχαριστώ πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφορία. Σας ευχαριστώ ε, για την παρέμβασή σας ε, και νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει και την εισηγητρία κατά την επανεξέταση του θέματος ως Επιτροπή. Θα βρούμε διατύπωση και απέναντι στους αναφέροντες όταν φτάσει η ώρα. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ χρήσιμο. Ας προχωρήσουμε τώρα, δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο για το συγκεκριμένο θέμα. Και γι' αυτό θα ήθελα να ενημερώσω όλους ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ε, σχετικά με τις συστάσεις της έκθεσης αυτής ε, είναι η 18η Οκτωβρίου, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, στις 3 η ώρα το απόγευμα. Ε, και η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου στην επόμενη δηλαδή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ε, Τζούντ, θα ήθελες να ξαναπάρεις το λόγο? Έχουμε χρόνο. Απλά θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συναδέρφους ε, για το συναδελφικό πνεύμα που επέδειξαν. Όπως είπες και εσύ, Σεσίλια, είναι πολύ λεπτό το θέμα και είναι δύσκολο και πολύ φορτισμένο θέμα. Και όπως είπα στο τέλος ε, της εισαγωγής μου, θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου τις μητέρες, τους πατέρες, τα αδέρφια που συναντήσαμε στη Μαδρίτη και που έχουν ε, παρουσιάσει τις αναφορές τους εδώ στην Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε απαντήσεις για αυτούς ε, σχετικά με το τι απέγιναν τα μέλη της οικογένειάς τους. Θα πρέπει λοιπόν ε, να τους υποστηρίξουμε όσο γίνεται και να φτάσουμε στην ψηφοφορία και μια καλή έκθεση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και σε ευχαριστώ για όλη τη δουλειά που κάνεις ε, στο δύσκολο αυτό θέμα. Να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Νομίζω ότι ήδη έχουμε εδώ τους αναφέροντες ε, για την αναφορά 1525. Είναι όλοι παρόντες. Καλώς ήρθατε. Θα εξετάσουμε λοιπόν τις ε, υποθέσεις ανεξιχνίας των ε, δολοφονιών ε, από την τρομοκρατική ομάδα ΕΤΑ στην Ισπανία. Καλωσορίζω όλους τους αναφέροντες και πολύ ευχαριστώ θα σας δώσω το λόγο. Καταρχάς, στον κύριο Ροδρίγες Αρίας και τον κύριο Πορτέρο Ντελατόρε. Πέντε λεπτά ο καθένας και κατόπιν θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τις ευρωβουλευτές και πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Sí. Καλησπέρα σα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές της ε, Επιτροπής, η Ένωση Αξιοπρέπεια και Δικαιοσύνη εμφανίζεται εδώ σήμερα γιατί 379 από τις 864 δολοφονίες ε, που διέπραξε η τρομοκρατική οργάνωση ΕΤΑ στην Ισπανία και στη Γαλλία εξακολουθούν να μην έχουν επιληθεί. Πρόκειται για περίπου ε, τις μισές. Μία στις δύο δολοφονίες της ΕΤΑ που έγιναν στην Ισπανία και στη Γαλλία, ένα 44%, ε, ακόμα και σήμερα δεν έχουν επιληθεί. Πρόκειται για 379 οικογένειες που συνεχίζουν χωρίς το θεμελιώδες δικαίωμα στη δικαιοσύνη και χωρίς να γνωρίζουν την αλήθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Χωρίς ε, αποτελεσματική δικαστική προστασία ε, για όλες αυτές τις ε, δολοφονίες, κάτι που αντιβαίνει στα άρθρα 2 και 47 της Ευρωπαϊκής Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα αρκετών ανώμαλων περιπτώσεων που ε, αντιβαίνουν στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης. Η, πρώτη είναι η σαφής παράβλεψη της εφαρμογής από πλευράς ισπανικών αρχών και της ε, ε, δικαιοσύνης ε, τη νομολογία που αναγνωρίζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας και από τον ποινικό κώδικα της Ισπανίας που επιτρέπει να δικαστούν οι επικεφαλεί της ΕΤΑ ε, που ήταν στα ενία κάθε φορά που διεπράχθηκε κάθε μία από αυτές τις 379 δολοφονίες. Αναφερόμαστε στο δόγμα της οργανιζιάς ΣΕΡΣΑΦ, ναι, της αρμόδιας αρχής που πρότεινε ο καθηγητής ε, Κλάους Ρόξιν από τη Γερμανία στα μέσα του προηγούμενου αιώνα και ε, την έχουν αναγνωρίσει και το Ανώτατο Δικαστήριο της Γερμανίας και το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας και έτσι επιτρέπεται ε, να λάβει κανείς δράση κατά των πραγματικών, των αυθεντικών δραστών, κατά των ανθρώπων που βρίσκονταν πίσω από τη δολοφονία. Αυτοί που ε, διέταξαν τη δολοφονία αυτών των ε, ανθρώπων. Το κράτος δικαίου έχει δικαίωμα να ε, στραφεί κατά όλων των δραστών, εκείνων που προετοίμασαν τις ε, βόμβες ε, που πάτησαν τη σκανδάλη αλλά και εναντίον όλων εκείνων οι οποίοι ήταν στα ενία της οργάνωσης ε, και που διέταξαν αυτούς τους δολοφόνους. Επιπλέον η Ισπανική αστυνομία και η Guardia Civil μπόρεσαν να γνωρίσουν ποιοι ήταν αυτοί οι επικεφαλείς της τρομοκρατικής οργάνωσης και το γνώριζαν ανα πάσα στιγμή. Και Γι' αυτό ακριβώς ε, θα θέλαμε να σας ε, προσκομίσουμε ένα ακόμα έγγραφο που είναι μια έκθεση η οποία αναφέρει όλους εκείνους τους επικεφαλείς που είχε η τρομοκρατική οργάνωση της ΕΤΑ έναν έναν. Ε, επιπλέον δε η δικαιοσύνη σε καμία περίπτωση δεν ξεκίνησε ερευνητικές διαδικασίες κατά οποιονδήποτε εκτός εξ αυτών των επικεφαλής δεν είναι ίση ενώπιον του νόμου αυτοί οι 379 δολοφονηθέντες βάσει ε, του άρθρου 20 ε, και 21 της Χάρτας των Θεμελών Δικαιωμάτων. Δεν έχουν ίδια δικαιώματα οι Ευρωπαίοι πολίτες βάσει του άρθρου 47. Δεν είναι εγγύηση και κατάλληλη προστασία μέσω της διαμεσολάβησης και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας στο δικαίωμα στη ζωή του άρθρου 2 στη, της Χάρτας, ο πυρήνας και μία από τις βασικές υποχρεώσεις όλων των κρατών μελών ε, για όλους τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, μπορούμε να αποδείξουμε ότι πέραν των όσων είπαμε παραπάνω, το Ισπανικό κράτος απέτυχε και στην έρευνα, ε, στην πραγματική και αποτελεσματική έρευνα αυτών των 379 υποθέσεων λόγω παραλήψεων, αμέλειας, ε, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι κατέστρεψαν μόνοι τους κάποια από τα αποδεικτικά στοιχεία της έρευνας. Και αποδείχθηκε αυτό με στοιχεία και σήμερα σας έχουμε φέρει ε, ένα νέο έγγραφο το οποίο το πιστοποιεί αυτό. Υπάρχει ένα επίσημο πιστοπιστικό από τις Ισπανικές Δικαστικές Αρχές που αποδεικνύει ότι η καταστροφή αυτών των αποδεικτικών στοιχείων είναι μία από τις 379 ε, θέσεις. Υπάρχει συγκεκριμένος όρος στην Ισπανία και υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και εδώ σας φέρνουμε τη, τα στοιχεία ενός εκ των θυμάτων. Επίσης υπάρχουν ε, ε, αντίστοιχες περιπτώσεις που αφορούν 379 δολοφονίες. Ολοκληρώνω. Ζητάμε όλα αυτά να διερευνηθούν. Γι' αυτό ακριβώς και σας ζητούμε να εξετάσετε την διερεύνηση όλων αυτών των υποθέσεων καταρχάς και να έρθει και μια αποστολή ευρωβουλευτών στην Ισπανία για να συναντηθεί με τα θύματα, με τις αρχές ε, ε, όπως έγινε πρόσφατα από την Επιτροπή σας και μάλιστα και σήμερα συζητήθηκε ε, για μια άλλη ανώμαλη δικαστική υπόθεση, αυτή η υπόθεση της ε, απαγωγής ε, των παιδιών, των stolen babies. Μην αφήσετε λοιπόν να ξεχαστούν στη λύθη αυτοί οι 379 πολίτες που δολοφονήθηκαν με τέσο βίαιο τρόπο και η οικογένειά τους. Θα πρέπει να σας διηγηθώ το εξής. Σήμερα είμαστε μια ομάδα θυμάτων εδώ, θυμάτων τρομοκρατίας, από τους οποίους έχουμε τέσσερις οικογένειες που σήμερα Εδώ στα μια αίθουσα σας παρουσίασαν πώς ε, δεν είναι δυνατόν να επιληθούν οι καταστάσεις τους, το γεγονός ότι δεν, υπήρξε, δεν αποδόθηκε δικοσύνη, ε, υπάρχουν ε, οικογένειες, εγώ είμαι θύμα της τρομοκρατίας, ο πατέρας μου δολοφονήθηκε το 2000. Εγώ είμαι θύμα της τρομοκρατίας, δολοφονήθηκε το 2000 ο πατέρας μου, αλλά εγώ δικαιώθηκα, ε, υπήρξε καταδίκη. Αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι άνθρωποι, άλλα θύματα της τρομοκρατίας που βρίσκονται εδώ σήμερα παρόντες και δεν είχαν την τύχη που είχα εγώ. Και το μόνο το οποίο ζητάμε είναι πραγματικά το Ισπανικό κράτος βάσει της Χάρτας των Θεμολογιών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει δράση. Και τώρα θα δώσω το λόγο σε ένα εξ αυτών των ανθρώπων Λοιπόν, για να σας περιγράψει την ε, κατάσταση ακριβώς. Ο Ίνικο Πασκουάλ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία να ακουστούν και οι φωνές των θυμάτων που είναι εδώ σήμερα. Το 1982 ο πατέρας μου Ήταν η τρίτη επιστολή αυτή που κατήχε και που του είχε στείλει η ΕΤΑ και στην οποία του έλεγε ότι αν δεν εγκατέλειπε την εργασία του ως διευθυντής της ε, κατασκευής του εργοταξίου ε, για την ε, μονάδα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας θα έχανε τη ζωή του. και μετά από λίγο καιρό δολοφονήθηκε από ένα συνεργάτη του με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Ο πατέρας μου με ρώτησε «Εσύ Ινίγον τι θα έκανες» και εγώ του είπα «Εσύ τι θα κάνεις» και λέει «Ε, ε, κανονικά θα έπρεπε να εγκαταλείψω τη θέση μου. Αλλά εγώ δεν θα το κάνω, δεν θα αφήσω τη θέση μου. Και δεν θα το κάνω για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί πιστεύω ακράδαντα σε αυτό που κάνω. Και ο δεύτερος διότι χρειάστηκα πολύ κόπο για να καταλήξω μέχρι εδώ. Όπως ε, ε σας είπα μερικές εβδομάδες αργότερα κάποιοι τρομοκράτες της ΕΤΑ, τέσσερις στον αριθμό, κατέβηκαν από έναν αυτοκίνητο και του έριξαν πάνω από 25 σφαίρες. Ήταν 8 το πρωί ε, της 5ης Μαΐου και το ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί ήμουν εκεί μαζί του. Μου στήχησε πάρα πολύ. Δυσκολεύτηκα να ανέβω πάνω στο σπίτι και να το διοικηθώ στη μητέρα μου και στις αδερφές μου. Μου στήχησε πάρα πολύ να τον αφήσω εκεί ε, από αυτό το αυτοκίνητο με όλες αυτές τις ε, σφαίρες. Λίγες ώρες αργότερα ήρθε αστυνομία στο σπίτι μου και μου είπαν, ε, με έκαναν πάνω από 100 ερωτήσεις, ε, μου έδειξαν πάνω από 100 φωτογραφίες ε, φερόμενων τρομοκρατών για να αναγνωρίσω ίσως κάποιον και θυμάμαι ότι μου είπαν μην ανησυχείς Ίνιγκο, θα τους πιάσουμε αυτούς τους δολοφόνους και θα τους βάλουμε στη φυλακή. 35 χρόνια μετά, ακόμα και σήμερα, Ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι δολοφόνησαν τον πατέρα μου και φυσικά δεν είναι και κανείς στη φυλακή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω γιατί τίνατε βίκονους αυτά που είχαμε να σας πούμε. Δυστυχώς ε, δεν μπόρεσαν να μιλήσουν όλοι, λόγω έλλειψη χρόνου μιλώ εγώ, αλλά υπάρχουν και άλλοι ε, συνάδελφοι που σκοτώθηκαν οι γονείς τους ε, στη δεκαετία του 70 και υπάρχουν και άλλοι ακόμα και πολλές υποθέσεις δεν έχουν επιληθεί. Εγώ νιώθω βαθιά Ευρωπαίος, πολύ πιο Ευρωπαίος από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί ο καθής και αυτό πολύ πριν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ισπανία. Γι' αυτό ακριβώς σας εκλυπαρώ να μας βοηθήσετε να καταπολεμήσουμε αυτή την ατιμορρησία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστώ για τη δήλωση την οποία κάναμε. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική και το ιδιαίτερα πάρα πολύ ανησυχητική. Πράγματι στραφήκατε σε εμά όχι σαν πολιτικοί αλλά σαν άνθρωποι και το εκτιμούμε αυτό. Και βλέπω και εγώ όλους τους συναδέλφους εδώ ότι έχουν συγκινηθεί από την δική σας ιστορία. Δεν είστε μόνος και από ό,τι φαίνεται υπάρχει κάποιο πνεύμα ατιμορρησίας πολιτιστικής το οποίο πρέπει να καταπολεμήσουμε. Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ομιλητές και συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Πριν ξεκινήσει όμως η συζήτηση, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά ας προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη την ιστορία την οποία ακούσαμε όχι να προσπαθήσουμε να επιτεθούμε ο ένας τον άλλο, αλλά να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα αιτήματα των αναφερόντων που έχασαν τους δικούς τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, συζητάμε εδώ μια σειρά ανεξιχνίας των υποθέσεων και η αναφέροντες βοηθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, ε, να αναλάβει δικαιοσύνη τους ανθρώπους αυτούς. Το εάν κάποιος είναι αθώος ή ένοχος ενός εγκλήματος ε, είναι ε, αρμοδιότητα αποκλειστικά του των εθνικών ε, κυβερνήσεων. Ε, αυτό απορρέει από το άρθρο 72 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Κατά αναλογία και καταλαβαίνω ότι αυτό δεν θα αρέσει στους ε, αναφέροντες. Ε, τα, όργανα της, ε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στην δικαιοσύνη των κρατών μελών. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με τα θύματα τρομοκρατίας. Ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να αυξήσουμε τα δικαιώματα των θυμάτων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει οδηγία το 2004 για την αποζημίωση και 2012 για τα δικαιώματα των ε, θυμάτων ε, και φέτος ε, έχει οθετήσει και την οδηγία κατά της τρομοκρατίας ε, που προβλέπει ειδική έκθεση αμέσως μετά την επίθεση και για όσο χρειάζεται κατόπιν. Και εμείς θέλουμε να δούμε εφαρμογή της οδηγίας αυτής μέχρι το Σεπτέμβριο του χρόνου. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται για την προστασία των θυμάτων της τρομοκρατία και εξετάζουμε και πιθανά περαιτέρω μέτρα. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ και να επισημάνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν λίγες μόλις εβδομάδες έλαβε απόφαση να ε, δημιουργήσει μια ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όλοι λοιπόν καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες. Αυτό δεν θα σας ε, φέρει πίσω τους ε, αγαπημένους σας ανθρώπους που χάσατε, αλλά θα μας βοηθήσει ε, να προστατεύσουμε ανθρώπους σε μελλοντικές περιπτώσεις. Ωραία, σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο πρώτα στους ευρωβουλευτές και μετά στους αναπληρωτές. Καταρχάς η κυρία Μπεατρής Πεσταίρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλώς ορίσατε όλοι όσοι είστε εδώ οι αναφέρονται στα θύματα και να ευχαριστήσω και τα μέλη που είναι επίσης εδώ ε, διότι ευτυχώς εδώ και μήνες που συζητούσαμε κατά πόσον θα παραμείνει ανοιχτή αναφορά και θα συζητηθεί εδώ στην Επιτροπή, ε, καταλήξαμε να, σε μια συμφωνία. Σε μια συμφωνία δικαιοσύνης και κοινή λογικής. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Ρώσα Εσταράς ε, για την υποστήριξη για την ε, αποφασιστικότητα και την επιμονή της, διότι πρέπει τουλάχιστον να ακούσουμε, να είμαστε σε θέση ε, να ε, ασκήσουμε πλήρως το δικαίωμα ε, που προέρχεται από αυτές τις αναφορές. Το θέμα της τρομοκρατίας στην Ευρώπη και τελευταία το νιώθουμε όλο και περισσότερο και ορισμένες φορές είναι όλο ένα και πιο σαφές ότι το να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και να συλλάβουμε τους υπόπτους σημαίνει ότι έχουμε και ευθύνη ενώπιον των θυμάτων και είναι ηθική υποχρέωση των χωρών μας ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να λύσουμε λοιπόν αυτά τα 400 περίπου εγκλήματα είναι υποχρέωση και για τα θύματα που βρίσκονται εδώ και για αυτούς που εκπροσωπούν. Πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν ε, ε, τις ανάγκες του, αλλά αυτό σημαίνει ότι στέλνουμε και μήνυμα στους τρομοκράτες για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση, προσπαθούν να καταστρέψουν τη δημοκρατία αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά αυτό σημαίνει και ότι τηρούμε και τι νομικέ υποχρεώσει Ευρωπαϊκή Ένωση και του διεθνού δικαίου. Και εγώ θα ήθελα με κάθε σεβασμό να ε, αποστείλω ένα μήνυμα ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση που μας έκανε και που μας είπε ότι πρόκειται απλώς για καθορισμό της αρμοδιότητας για το κατά πόσον θα υπάρξει μια ε, επίλυση της υπόθεσης. Ναι, αλλά εδώ δεν λέμε απλώς ε, ότι αναφέρονται ζητούν να επιληθεί ένα ποινικό ζήτημα. Αναφέρονται στα δικαιώματα των θυμάτων και δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε και αυτό το να σταματήσει η ατιμορρησία, να μάθουν ποιοι ε, σκότωσαν τους ε, ε, συγγενείς τους είναι δικαίωμα. Είναι δικαίωμα όπως όλα τα υπόλοιπα. Είναι βασικό δικαίωμα και ως βασικό δικαίωμα που περιλαμβάνεται στη Χάρτα των Θεμελωδών Δικαιωμάτων είναι τμήμα των υποχρεώσεών μας ως θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε την κατάσταση των εγκλημάτων που διέπραξε η ΕΤΑ, κυρίως διότι όπως είπε και εσείς με τη νέα οδική για την τρομοκρατία όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πώς μπορεί ένα τόσο μεγάλο αριθμό ε, αριθμός ε, ε, δολοφονιών δεν έχει ακόμα επιληθεί. Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει και κοινωνικές επιπτώσεις και πρέπει να προστατεύσουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πολιτικά δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να ζητήσω να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά διότι θεωρώ ότι πρέπει να αποστείλουμε ε, μία επιστολή στη Νέα Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξηγήσουμε και να ζητήσουμε τη συμμετοχή τους ε, για την όλη διαδικασία και επίσης θα ήθελα να ζητήσω να σταλεί και επιστολή στην κυβέρνηση της Ισπανίας. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ε, είναι βαθύτατα εμπλεκμένη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάψει η ατιμορρησία και να πάψουν να υποφέρουν τα θύματα. Θύματα στα οποία οφείλουμε κάθε σεβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μπεατρίθ. Ρώσα. Η κυρία Σταράς παγραγούτ Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για την παρουσία τους εδώ όλους τους εκπροσώπους των θυμάτων που είναι μαζί μας σήμερα. Πραγματι υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με το ότι δεν έχουν καταλήξει οι υποθέσεις για τα μισά τουλάχιστον από τα εγκλήματα στα οποία προχώρησε η ΕΤΑ. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, 397 εγκλήματα, το 44% είναι ανεπίλητα και ζήτησαν πλέον να έρθουν εδώ για να δικαιωθούν. Η απάνταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θυμίζει τη στάση που κράτησε και στην επίσκεψη που είχαμε κάνει στην Ισπανία για τα, τις απαγωγές των παιδιών. Είπε ότι δεν είναι αρμόδια. Εμείς εμένουμε όμως ότι είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν πρώτη ανησυχία έχει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα λοιπόν είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όπως είπαμε και στην περίπτωση των απαγωγών, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμπλακεί, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να βοηθήσει τις προσπάθειες που κάνουν τα θύματα, να βοηθήσει την Ισπανική κυβέρνηση, να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να διελευκάνουμε κάθε μία από τις δολοφονίες αυτές. Γι' αυτό λοιπόν ζητείτε η βοήθεια της ε, Επιτροπής να υπάρξει και μία, εγώ στηρίζω την πρόταση για να υπάρξει μία επίσκεψη διερευνητική στην Ισπανία. Είναι αλήθεια ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι στην ουσία ένα μέσο πίεσης. Δεν μπορούν να μιλήσουν όλοι, υπάρχουν όμως μαρτυρίες ε, μια συντρόφου που σκότωσαν τους ε, συγγενείς της, τους θείους της και μάλιστα σε μια περίπτωση ήταν και η τελευταία θανατηφόρα επίθεση της ε, οργάνωσης ΣΕΤΑ Υπάρχουν πολλές μορφές θυμάτων λοιπόν της τρομοκρατίας. Θα είναι αλήθεια ότι το θέμα της επίλυσης των θεμάτων αυτών, των δολοφονιών αυτών, είναι θέμα πριν από όλα δικαιοσύνης. Η πρόεδρός μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί ιδιαίτερα και, σαν, και ιδιαίτερα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν μπορεί να, μην κάνει, να κάνει παρά ό,τι περνάει από το χέρι της η Επιτροπή μας έτσι ώστε να επιληθούν όλες αυτές οι περιπτώσεις να στείλουμε επιστολές και στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας από πλευρά της Ισπανικής κυβέρνησης έτσι ώστε επιτέλους να βρεθεί μια λύση σε, όλα αυτά τα, όλες αυτές, για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ κύριος Λόπες Αγουιλάρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Για, για μια ακόμη φορά θέλω να χαιρετήσω εδώ όλους τους ε, εκπροσώπους των οργανώσεων των θυμάτων και των αντιτρομοκρατικών οργανώσεων. Ε, φυσικά η περίπτωση της Ισπανίας ε, είναι μια πολύ διαφωτιστική περίπτωση. Ε, πράγματι είναι, είμαστε μια περίπτωση η οποία έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον. Δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει με αυτά τα οποία ακούσαμε θα ήθελα να χαιρετήσω προσωπικά όλα τα θύματα που είναι εδώ και τους εκπροσώπους των θυμάτων και θα πρέπει όλα τα δημοκρατικά κόμματα όχι μόνο να ενωθούμε σε σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αλλά να πάρουμε κάθε μέτρο το οποίο είναι απαραίτητο για να υπάρξει ένα τέλος στις τρομοκρατικές δραστηριότητες για να υπάρξει επιτέλους απόδοση δικαιοσύνης γιατί όπως είπαμε 379 δολοφονίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν διελευκανθεί και υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες επίσης οι οποίες ζητούν να υπάρξει αποκατάσταση και δικαιοσύνη. ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να είναι αρμόδια ε, λόγω της νομοθεσίας αλλά θα πρέπει να ακούμε, θα πρέπει να ακούμε με ευαισθησία και να προσπαθήσουμε να δούμε ε, τι μπορούμε να κάνουμε γιατί πράγματι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με δική του πρωτοβουλία έχει κάποια μέσα τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί και ε, να προσπαθήσουμε ε, και στα πλαίσια της οδηγίας για την προστασία των θυμάτων του 2012 όπως επίσης και των θυμάτων της τρομοκρατίας του 2007 να εξαντλήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να βρεθεί μια λύση. Νομίζω ότι η εμπειρία της Ισπανίας και της ενότητας των μεγάλων δημοκρατικών κομμάτων ήταν αποφασιστική έτσι ώστε να κινητοποιηθεί η δικαιοσύνη, να, να κινητοποιηθεί η εισαγγελία και όλες οι οργανώσεις οι δικαστικές έτσι ώστε να τεθεί ένα τέλος στις δραστηριότητες της ΕΤΑ ολοκληρώθηκε ένα τμήμα της ε, υπόθεσης αυτής, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει πάντα το θέμα αυτό για το οποίο είναι σήμερα εδώ ε, τα θύματα, ή εκπρόσωποι των θεμάτων. Ε, το θέμα αυτό θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό σε συζήτηση, θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Ακούσαμε με πόσο συναισθηματικό τρόπο αλλά και αξιοπρέπει την σημασία που έχει αυτό το θέμα. Λοιπόν, θέλω να να πω ότι εμείς αποτείουμε φόρο στα θύματα της θερμοκρατίας και τους Ισπανούς σε όλους αυτούς ε, που καταπολέμησαν την ΕΤΑ. Εγώ έχω γνωρίσει πάρα πολλούς που πολέμησαν εναντίον της τρομοκρατίας και έπεσαν θύματα και μπόρεσα να εκτιμήσω ακριβώς ότι είχε κάνει και ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδα γύρω από αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχατε μάλιστα την ευκαιρία να γνωρίσετε τον πατέρα του. Η Βρυξέλλες είναι το μέρος όπου συναντιέται ο κόσμος. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι τόσες ε, ελπίδες ε, γεννιούνται στις Βρυξέλλες εδώ αυτή τη στιγμή και όλα σε τούτη την αίθουσα. Ο κύριος Διάστεμερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχετε πολύ ωραία μάτια, αλλά σήμερα είναι δακρυσμένα και πραγματικά είναι βουρκωμένα όπως και τα μάτια της Ρώσα. Η αρμοδιότητα της Επιτροπής, ε, κατά την άποψή μου, είναι αδιαφυσβήτητη. Πρόκειται για μια πολιτική επιτροπή, η οποία έχει πολύ μεγάλη πολιτική ισχύ. Και αναφερόμαστε εδώ σε 379 θύματα, στα οποία δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, δεν έχουν αποζημιωθεί και δεν έχουν παρηγοριά και είναι κοινή λογική ότι η ατιμορρησία αποδυναμώνει το δίκαιο και ενισχύει το δολοφόνο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να κάνω επίκληση ε, σε πολιτικό επίπεδο για την ελληνική αυτής της Επιτροπής. Την ε, δύναμη που έχει στα μέσα η Επιτροπή, την ε, απαραίτητη συμπάθεια και συμπαράσταση αυτής της Επιτροπής. Η δέσμευσή σου, Σέιλια, την οποία έχουμε αναγνωρίσει πάρα πολλές φορές, ε, διότι είσαι στρατευμένη στην υπεράσπιση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εισαγγελία και η ε, ισπανική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητες. Δεν συμφωνώ με το σχόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το άρθρο 77, 72, συγγνώμη, την αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ήδη γνωρίζουμε ποια είναι η αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αλλά γνωρίζουμε επίσης και ποια είναι η πολιτική ισχύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σίγουρα αυτή της Επιτροπής. Εάν οι φίλοι μας που είναι εδώ σήμερα κάθονται πίσω στους οποίους θα ήθελα να ε, εκφράσω το θαυμασμό, το σεβασμό και την αλληλεγγύη μου. Αν συμφωνούν λοιπόν, ε, ό,τι μας πούν αυτοί, αν συμφωνούν λοιπόν, τα έργανα της Επιτροπής μπορούν να αποτανθούν στην ε, ανεξάρτητη εξουσία της Αγγελίας και της Δικαιοσύνης της Ισπανίας και στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η Ντολόρες Δελγάδο είναι μια πολύ ικανή εισαγγελέα, αρμόδια για το συντονισμό της ε, καταπολέμησης ε, της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας και γνωρίζει για τον πόνο των θυμάτων. Ας γράψει η Επιτροπή στην Ντολόρες. Ο Γενικός Εισαγγελέας του κράτους ε, επίσης είναι κάποιος τον οποίο μπορείτε να γράψετε. Ε, τον, ε, στον εισαγγελέα επίση ε, της Εθνικής Συνέλευσης και σε αυτόν μπορείτε να γράψετε. Μπορείτε να γράψετε επίση και στον πρόεδρο του Εθνικού Δικαστηρίου και μπορείτε να γράψετε και στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τίποτα άλλο και ευχαριστώ πολύ. Γράφω τόσο γρήγορα και ζητήστε, σας ζητώ συγγνώμη που καθυστερώ λίγο να απαντήσω. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Μάιτε. Το επίθετό σας είναι τόσο δύσκολο που δεν τολμώ καν να το προφέρω. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω πολύ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να σας πω μια ιστορία πέντε χρόνια ε, τρεις μεγάλοι ε, ερευνητέ ε, συνέλεξαν στοιχεία όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας και της ΕΤΑ και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων και μπόρεσε να δημοσιευθεί αυτό το βιβλίο για πρώτη φορά. Το 2010. Μόνο όταν δημοσιεύθηκε αυτό το βιβλίο, εκδόθηκε το βιβλίο, ένα άτομο που γνωρίζουμε πολύ καλά, ο Ντάνι Πορτέρο και εγώ, ο ε, Δελγάδο κατάλαβα ότι έπρεπε να επιληθούν πάνω από 3.000 υποθέσεις και εκκρεμούν 379. Αναφερόμαστε στο 2010. Μιλήσαμε και με τον επικεφαλής ε, του ε, Αθηνικού Δικαστηρίου και του δώσαμε προσωρινά αυτά τα στοιχεία και μας είπε είναι αδύνατο. Για 1,5 χρόνο δίναμε μάχη για να εξακριβωθούν τα στοιχεία και είναι ακριβή. Το 2010 αυτό. Και υπάρχουν υποθέσεις ε, σαν τον ε, κύριο του Κοράλ και άλλους φίλους που ε, τους ε, σκότωσαν στην Γαλλία όταν πήγανε να δουν μια ταινία και ήταν δικτατορία ακόμα και τότε δεν τους επέτρεπαν να δουν κάποιες ταινίες. Τους θεώρησαν αστυνομικούν και τους ακροτηρίασαν, τους βασάνισαν μέχρι που τους δολοφόνησαν. Το ξέρουμε, υπάρχουν άνθρωποι που τα μαστά ε, περιέγραψαν, αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ τα σώματά τους. Οι οικογένειές τους δεν μπόρεσαν να αντέξουν τον πόνο και αυτό είναι θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να βρούμε τις νομικές οδούς, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βοηθήσουμε. Τώρα που ε, αντιμετωπίζουμε, κλείνει το θέμα της ε, τρομοκρατίας στην Ισπανία, έχουν εκατοντάδες δολοφονίες στους δρόμους και δεν υπάρχει δικαιοσύνη και είναι αδύνατο να ε, τιμήσουμε και τη μνήμη αυτών των θυμάτων. Έχουμε εκατοντάδες υποθέσεις ανεπίλητες και πραγματικά αυτοί που έχουμε ζήσει τον δρόμο της δολοφονίας στον περίγυρό μας αλλά έχουμε δικαιωθεί ήταν πάρα πολύ μεγάλη η ανταμοιβή. Ε, αυτός ο, ο, ο τρόμος χωρίς να δικαιώνονται αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους βλέπουμε εδώ σήμερα, αξίζει την προσπάθεια όλων. Αξίζει την προσπάθεια όλων εδώ στην ε, Επιτροπή. Αξίζει να αναζητήσουμε, να προσπαθήσουμε, ώστε ό,τι είναι δυνατό και να μπορέσει να τους δικαιώσει με κάποιο τρόπο, να τους δοθεί. Σας εκλυπαρώ λοιπόν να λάβετε υπόψη σας όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι 8 χρόνια σε αυτό το κοινοβούλιο και όπως η ΜΑΙΤΕ και όπως ο προηγούμενος συνάδελφος Είχαμε θύματα και τα ονόματα των θυμάτων αυτών βρίσκονται μέσα σε αυτό το βιβλίο και από 8-9 ετών μετά τη δολοφονία του Αλμπέρτο κάποιοι από τους δολοφόνους καταδικάστηκαν. Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται στη φυλακή. δεν είχαν όλη την τύχη την οποία είχα εγώ σε σχέση με την καταδίκη των δολοφόνων μετά από τον φόνο του αδελφού μου. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να έχουν και αυτοί ε, την ίδια τύχη την οποία έχω εγώ και να δουν αυτούς οι οποίοι εκτέλεσαν τα εγκλήματα αυτά στη φυλακή. Υπάρχουν λοιπόν 379 ε, νέκροι των οποίων ε, οι υποθέσεις δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα πλήρως και δεν έχουν επιληθεί. Θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατό από αυτό το κοινοβούλιο έτσι ώστε να καταδικαστούν αυτοί που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα. Τα εγκλήματα αυτά είναι εγκλήματα εις βάρος της ανθρωπότητας. Είναι η μοναδική ευκαιρία την οποία έχουμε να το κάνουμε αυτό αν δεν θέλουμε κάποτε να παραγραφούν. Είναι νόμιμο δικαίωμα, θεμητό ε, να ζητήσουμε να υπάρξει πραγματική ε, δικαίωση. Αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη είναι και το όνομα μίας από τις οργανώσεις που εκπροσωπούνται εδώ σήμερα αυτό το οποίο ένα πράγμα είναι που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η γραπτή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγει το εξής ότι η οργάνωση αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη ανησυχεί να παραπέμψει τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη ε, και όχι τόσο να προστατεύσει τα δικαιώματα των θυμάτων της τρομοκρατίας. Αυτός ο οποίος το έγραψε αυτό δεν γνωρίζει τα πραγματικά θύματα της τρομοκρατίας, δεν έχει μιλήσει μαζί τους και δεν ξέρει ότι το πραγματικό που παίζει ρόλο, που μετράει είναι η αλήθεια, η δικαιοσύνη ε, και είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε την συγκεκριμένη αναφορά ανοιχτή είναι σαφές ότι ανήκει στις αρμοδιότητές μας, είναι κάτι το οποίο άπτεται και του κεφαλαίου 6 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να κλείσουμε την υπόθεση αυτή. Μιλάμε για το τέλος της ΕΤΑ, μιλάμε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και της ειρήνης αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη όχι μόνο για την ΕΤΑ, για την Κολομβία κτλ. που να μην βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης. Αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη. Γιατί αυτά τα θύμ, πώς μπορούμε εμείς να μιλήσουμε για την ΙΤΑ και την καταστροφή της ΕΤΑ όταν έχουμε τα θύματα αυτά εδώ σήμερα. Ναι με να κατησχίσαμε σε επίπεδο στρατιωτικό ή αστυνομικό, αλλά όταν υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ δεν έχει υπάρξει πραγματική δικαιοσύνη. Εμένα δεν έχει σημασία το ότι δολοφονήθηκε ο αδελφός μου. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι έρχονται από τη μία περιοχή ή την άλλη για να δολοφονήσουν τους αθώους. Λοιπόν, θα πρέπει να παραμείνει η συγκεκριμένη αναφορά ανοιχτή. Θα πρέπει να αποστείλουμε όλες τις επιστολές οι οποίες θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο. Γιατί όχι μόνο οι άνθρωποι αυτοί χάσανε και χάσαμε τους αγαπημένους μας, αλλά στην ουσία υπάρχει μια διπλή θυματοποίηση. Όχι γιατί μόνο δεν υπήρξε, υπήρξε η απώλεια των αγαπημένων μας, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει υπάρξει δικαιοσύνη, δεν υπήρξε απονομή δικαιοσύνης και σύν τις άλλες πολλές φορές δεν γνωρίζουμε καν πού είναι τα σώματα των ανθρώπων τους οποίους χάσαμε. Πρέπει λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη αναφορά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι πολύ ισχυρή αυτή η δήλωση και σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή. Συνήθως δεν έρχεστε. Το εκτιμώ ιδιαίτερα λοιπόν. Τώρα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Θηλουάγα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που πάντα μας δίνετε το λόγο στην Επιτροπή Αναφορών και ε, να ευχαριστήσω και τους αναφέροντες για τη σημερινή τους παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γιατί μας αφηγήθηκαν αυτή την ιστορία, ε, την τόσο προσωπική και τόσο γεμάτη πόνο. Οι αναφορές ε, που έστελναν και συζητιούνται εδώ στην Επιτροπή και στο αίτημα για ικανοποιητικές εξηγήσει προς την Ισπανική κυβέρνηση για τις δολοφονίες αυτές που δεν έχουν διαλευκανθεί και την ενημέρωση για την πρόοδο των ερευνών ε, μας φαίνονται ότι είναι καθόλου ε, λογικές και κατάλληλες και νομιμοποιούνται πλήρως. Δυστυχώς η κοινωνία μας εδώ και δεκαετίες έζησε με ε, φυσικό τρόπο την ε, βία ως μέσο για να επιτευθούν συγκεκριμένοι πολιτικοί στόχοι. Αυτό αδιαφυσβήτητα ήταν εσφάλμα και είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να εξαλείψουμε οριστικά από την κοινωνία μας. Ε, η βία της ΕΤΑ που είναι αυτή που συζητούμε σήμερα αλλά και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων και δυστυχώς και του κράτους σε κάποιες περιπτώσεις δεν ε, ε, έχει καμία δικαιολογία και φυσικά την απορρίπτουμε πλήρως, την καταδικάζουμε και θα έπρεπε να την καταδικάζουν όλοι. Ε, τα θύματα αυτών των εγκλημάτων που συζητούμε σήμερα ε, αξίζουν σίγουρα την αλληλεγγύη μας αλλά και επίσης την αναγνώριση και την ε, δυνατότητα της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Το δικαίωμα στην ε, αλήθεια και στην ε, ε, δικαιοσύνη, διότι αυτό είναι το δικαίωμα του καθενός και είναι και ικανή και αναγκαία συνθήκη για την αποκατάσταση της ειρήνης στην χώρα των Βάσκων, στην Ισπανία και φυσικά σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάω στον τελευταίο μιλητή στον κατάλογο, τον κύριο Κάλβε. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ε, ξεκίνησα στα αγγλικά, διότι άκουσα όλους ε, τους Ισπανούς ε, συναδέρφους και άλλους Ισπανούς να μιλούν Ισπανικά, αλλά μπορεί να φαίνεται ότι είναι αποκλειστικά Ισπανικό πρόβλημα. αλλά ως Ισπανικό πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Εγώ όμως βλέπω το θέμα ακόμη ευρύτερα, διότι μιλάμε για γενικές αξίες, ευρωπαϊκές αξίες και αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω. όσον αφορά την, ε, τη διοικητική νομική πλευρά μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην έχει αρμοδιότητες, αλλά η δική μας Επιτροπή Αναφορών έχει δικαίωμα και υποχρέωση να λάβει υπόψη το τι διακυβεύεται. Και αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η δικαιοσύνη. Η προστασία της δημοκρατίας από τη βία των εγκληματιών και αυτό είναι σημαντικό. Θα συνεχίσω στα ισπανικά αν μου επιτρέπετε. διότι θέλω να επιδείξω και αλληλεγγύη στα ε, θύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην επιτραπεί η τιμωρησία. να μην φαίνεται προφανέστατο ότι δεν γίνεται τα πάντα, γιατί αυτό πάλι ατιμορρησία είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ε, ο υποκινητής, ε, στον οποίο αναφέρθηκε η φίλη μου Τερέσα Χιμένες Πεχερίλ, ο υποκινητής, όχι ο εκτελεστής, αυτός που υποκίνησε το έγκλημα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Όχι. Ωραία. Και επιμένω ο υποκινητής, τον οποίο αναφέρθηκε η Τερέζα ε, Χιμένες Μπεθερίλ, όχι ο εκτελεστής, αλλά να υπάρχει δυνατότητα τη σήμερον ημέρα να το αναλάβει ε, κάποια ε, περιοχή της Ισπανίας γιατί δεν έγινε η απαραίτητη έρευνα. Και από εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος της ατιμορρησίας. Και φυσικά υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα. Και το λέω και το λέω μόνο στα ισπανικά. Γιατί πρέπει να παρεύει η Επιτροπή Αναφορών, γιατί πρέπει να κάνετε τα πάντα. Υποστηρίζω όλα όσα ακούστηκαν από τους συναδέλφους. Πρέπει να παρέμβει για ένα λόγο που θεωρώ ότι είναι απαραίτητος όσον αφορά τις αξίες Λυπάμαι για τους ε, φίλους, εγώ δεν, αντέχω σε κανένα, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, ανήκα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαι βέβαιο ότι δεν γίνεται ό,τι είναι δυνατόν. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια πολιτική ανοχής ε, με τους ε, συλληφθέντε πρώην εγκληματίε της ΣΕΤΑ. Υπάρχει μια πολιτική ανοχής που εμένα μου φαίνεται καλή μεν εκτός ενός πράγματος να απελευθέρωνονται χωρίς να υπάρχει απέτηση, χωρίς να υπάρχει απέτηση να συνεργαστούν ε, στη διαλεύκανση αυτών των δολοφονιών. Είναι ένα από τα πολλά που θα μπορούσαν να γίνουν. Το γεγονός όμως είναι ότι μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα και ε, ζητώ η Επιτροπή, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η Επιτροπή Αναφορών να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την υπόθεση και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πάντα η Επιτροπή αυτή ήταν στο πλευρό των θυμάτων ε, πέραν των νομικών και διοικητικών θεμάτων και να επιδείξω όλη μου την αλληλεγγύη και στις δύο συναδέλφους αλλά και σε όλους εκείνους που βρίσκονται στα πίσω έδρανα. Ευχαριστώ. Mr. Lopez White. Ο κύριος Λόπες is White. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα μιλώ ως Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διότι σήμερα Είχαμε και την ε, επέτειο του ε, πρώην ε, Προέδρου Βίλφρετ Μάρτιν και ήταν εκεί όλοι οι θύνοντες και καταφέραμε σήμερα μέσω εμού να σας διαβιβάσουμε σε όλους εσάς τα θύματα, τη στήριξη, τη στοργή και την αγάπη του ΕΛΚ. Κάθε φορά που συνεργαζόμαστε κερδίζουμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα όσα είπε ο συνάδελφος ο Χουάν Φερνάντο Λόπεθ Αγγιλάρ. Είναι αλήθεια ότι η ενότητα κατά τη ΣΕΤΑ ήταν και εξακολουθεί να είναι ε, ουσιαστική, ιδιαίτερα σε όργανα όπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το γεγονός ότι μας βλέπουν ενωμένου ε, εδώ σήμερα και ε, συναδέλφους από άλλες συνθέσεις, πολίτες, ανεξαρτήτους να μην αφήσουμε έξω κανέναν. Το γεγονός λοιπόν ότι είμαστε εδώ ε, Ευρωπαίοι σύντροφοι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα έτσι πρέπει να είναι. Εδώ και χρόνια, πριν γίνω Ευρωβουλευτής, ήμουνα βοηθός, δεν ξέρω ε, αν το ξέρουν οι συνάδελφοι, ότι έχω περάσει και κάποια χρόνια παραπάνω. Είμαι εδώ από τη δεκαετία του 90. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο τότε να εξηγήσουμε το φαινόμενο ΕΤΑ. Θεωρούνταν μια εξωτική τρομοκρατική οργάνωση, αποσχιστική, εθνικιστική και χρειάστηκε χρόνια για να εξηγήσουμε στους αδέλφους ότι πρόκειται απλώς για μια οργάνωση μαφιόζων δολοφόνων ενώ σκότωναν συντρόφους μας, σκότωναν ε, συγγενείς μας με υπομονή μέσω της του νόμου και μέσω του συντάγματος που είναι και η μάχη που πάντα πρέπει να δίνουμε στη χώρα μας σήμερα Είμαστε, όχι, δεν θα έλεγα σε τελείως διαφορετική εικόνα, ποτέ δεν πρέπει να ρίχνουμε τις αμυνέμες μας, γιατί το φαινόμενο επαναλαμβάνεται, εμφανίζεται με διαφορετική μορφή ο εθνικισμός, το μίσος, η προκατάληψη ε, σε κάποιες ε, περιοχές της Ισπανίας αλλά και σε ε, κάποιες περιοχές της Ευρώπης έχουν κάποιους παραλληλισμούς. Το μίσος για τη δημοκρατία και για τα όσα εμείς υπερασπιζόμαστε. Όλοι όσοι είμαστε εδώ νομίζω ότι συμφωνούμε από αυτού χωρίς καμία εξαίρεση θα ήθελα να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την επόμενη εβδομάδα έχω ένα γεύμα με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ζαν claude Juncker, και θα του σχολιάσω αυτήν την ε, ατυχή έκφραση, θα το πω διπλωματικά, που θα ήθελα να ζητήσω να διαγραφεί από το κείμενο. Λέει ότι αυτή ε, η Ένωση, η διγνητά η Χουστήθια, που όπως σχολίασε η συνάδελφος Τερέζα Χιμένες Μπεθερές, θέλει ε, να βρεθούν ενώπιον του δικαστηρίου άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με τρομοκρατικέ υποθέσεις. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα στην πρόθεση να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι ενώπιον του δικαστηρίου από ό,τι κατάλαβα ότι μπορεί να, μπορεί να υπήρχε και πρόβλημα μετάφρασης και ζήνω χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επανορθώσει αμέσως ή να ε, περιμένουν και τις πολιτικές συνέπειες για την υπόθεση αυτή. Θα το διαβιβάσω λοιπόν στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα όπως σας είπα. Και επίσης να πω και στα θύματα έχουν, ε, ακούσαμε εδώ σημερινέ ε, προσωπικέ αφηγήσει. Ε, κάποιοι από εμά έχουμε βιώσει διαφορετικέ συνθήκε, αλλά τίποτα, τίποτα δεν συγκρίνεται με το να σου στερούν ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Και θα ήθελα για άλλη μια φορά να επαναλάβω την υποστήριξη, την αλληλεγγύη, όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, αλλά όπω αποδείχθηκε, και αν είμαι και ο τελευταίο που μιλάω, θα ήθελα να το πω και σε όλου του συναδέλφου από όλα τα πολιτικά κόμματα, να σας ευχαριστήσω και ευχαριστώ και για τις ε, μαρτυρίες αυτές. Πάντα είναι απαραίτητο να έχουμε τέτοια πράγματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Thank you very much. And... Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει αμέσως σε αυτά τα οποία ακούστηκαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά. Προφανώς και εμείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή φροντίζουμε για τα θύματα της δημοκρατίας και δεν είπαμε ποτέ ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι. Υπήρξαν κάποια σχόλια από δύο ευρωβουλευτές για την πρώτη παράγραφο στην γραπτή απάντηση την οποία δώσαμε στο Κοινοβούλιο. Να προσπαθήσω να το εξηγήσω λίγο. Οι υπηρεσίες μας οι οποίες εργάζονται με τα θέματα καταπολέμησης ε, της ε, τρομοκρατίας και με τα θέματα ε, των δικαιωμάτων των θυμάτων της τρομοκρατίας και η οργάνωση αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη ασχολείται με τα θέματα των δικαιωμάτων των θυμάτων και κυρίως το θέμα της αναφοράς είναι τα 379 θύματα των οποίων οι υποθέσεις δεν έχουν ακόμα βρει μια λύση. Υπάρχουν δηλαδή δολοφονίες οι οποίες δεν έχουν διαλευκανθεί πάρα πολύ απλά. Δεν έχουμε πει κάτι το διαφορετικό από αυτό το οποίο μόλις είπα. Σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση αυτή. Για μια ακόμη φορά θα ήθελα να ζητήσω από τους ε, αναφέροντες να πάρουν πάρα πολύ ε, σύντομα το λόγο θα κάνουμε το ίδιο το οποίο κάναμε προηγουμένως. Έχετε το λόγο ε, για δύο λεπτά και εφόσον το επιθυμεί και ο επόμενος για δύο λεπτά επίσης. Ο κύριος Ροδίγες Αρίας πρώτος. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για, όλες τις, ε, για όλα τα δείγματα στήριξης τα οποία ακούσαμε εδώ Ακούσαμε ξεκάθαρες ιδέες, δεν ζητάμε εδώ για θέματα αθωότητας ή ενοχής. Λέμε ότι δεν έχει υπάρξει επαρκής έρευνα και αναζήτηση αυτών οι οποίοι είναι είτε αθώοι είτε ε, ένοχοι. Αν δεν υπάρχει σωστή ε, προσπάθεια έρευνας για την αλήθεια, δεν υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχουν και δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η βασική μας αρχή και έτσι θα στηρίξουμε ουσιαστικά τα θύματα. Να πω ότι είναι θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων. 379 οικογένειες, όχι μόνο οι δολοφονημένοι, πίσω από τα θύματα. Είναι 379 οικογένειες οι οποίες αναζητούν τη δικαιοσύνη και αναζητούν τον σεβασμό της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ζητάμε από την, Ευρωπαϊκή, από την Επιτροπή σας εδώ και χρόνια έχουμε θέσει το θέμα, έχουμε συναντήσει πάρα πολλά εμπόδια και παρακαλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προστατεύσει το δικαίωμα στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα ε, και τα δικαιώματα τα ανθρώπινα των θυμάτων αυτής της ε, ε, περίοδου. Ίσως είναι απαραίτητο να αποστείλετε μια, μια ομάδα στην Ισπανία μην αφήσετε τα θύματα αυτά μόνα τους. Εδώ και 40 χρόνια πολλά από αυτά είναι μόνα τους. So the other speaker left. Ο άλλος ομιλητή, αποχώρησε. Ο κύριος Πορτέρο Ντελατόρε. Έχετε κάτι να προσθέσετε. Ναι. Απλώς να πω, δεν ξέρω αν αυτό το οποίο σας αφηγήθηκε σας ράγισε την καρδιά ή όχι. Όλες οι απαντήσεις, όλες όμως οι απαντήσεις που άκουσα σήμερα από εσά ε, άγγιξαν τη δική μου την καρδιά. Εξ ονόματος των συναδέλφων μου και ε, δικού μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Σήμερα είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή εδώ στην Επιτροπή. Ε, σπάνια ακούμε και βλέπω και όλα τα μέλη να συμφωνούν με αυτή την άποψη ότι πρέπει πράγματι κάτι να γίνει. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι και αυτός νιώθει ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να κάνω είναι να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και να διαβάσουμε ένα μήνυμα σε αυτά τις 379 οικογένειες, τις ευρωπαϊκές οικογένειες που ακόμα περιμένουν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και επίσης θα ήθελα να διαβάσω και ένα μήνυμα πάθους και συμπόνιας για τα όσα αντιμετωπίζουν. Και μπορώ να το κάνω αυτό ως πρόεδρος της Επιτροπής εξ ονόματος όλων των μελών της Επιτροπής. Περιμένουν να αποδοθεί δικαιοσύνη και μέχρι σήμερα μάταια. Και πραγματικά θεωρώ και εγώ ότι αυτή η νοοτροπία της ατιμορροσίας πρέπει πλέον να σταματήσει. Ακούσαμε για τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, ότι επιθυμείτε να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα άρθρα. Μπορούμε να κάνουμε ελάχιστα, διότι εμείς δεν είμαστε δικαστική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά προσπαθούμε να βρούμε και λύσεις εξοδικαστικές σε ε, συνεχιζόμενες και μακροχρόνιες ε, διαφορές. Και αυτή σίγουρα είναι μια διαφορά που διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να με υποστηρίξουν οι συνάδελφοι στην πρότασή μου. Εννοείται ότι η αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή και θα τη στείλουμε στη νέα αρμόδια επιτροπή για την τρομοκρατία ε, προ ενημέρωση για να επιστήσουμε την προσοχή τους σε αυτή την υπόθεση η οποία διαρκεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και ε, διότι θα πρέπει να τη γνωρίζουν όταν εξετάζουν ε, αντίστοιχε υποθέσει και προετοιμάζονται για το μέλλον. Επίσης θα πρέπει να στείλουμε και ε, πλειάδα επιστολών ε, στις αρχές ε, στην Ισπανία, στο Γενικό Εισαγγελέα, στο Ανώτατο Δικαστήριο, στον Υπουργό Δικαιοσύνη, για να επισημάνουμε την κατάσταση, να πούμε ότι ακούσαμε τις υποθέσεις σας, ότι μάθαμε για το βιβλίο, για την ταινία και Κυρίως ακούσαμε τις προσωπικές σας ιστορίες και αυτό είναι τμήμα ε, του πόνου της Ευρώπης. Δεν είναι τοπικός, δεν είναι εθνικός, δεν είναι μόνο η οικογένειά σας. Ε, είναι μια ευρωπαϊκή πληγή ε, στην ευρωπαϊκή ανθρωπότητα και πραγματικά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Θα κάνουμε λοιπόν τα εξή και θα ζητήσουμε από όλου εκείνου που θα λάβουν αυτέ τι επιστολέ να κάνουν τι κατάλληλε έρευνε για αυτό το θέμα και να μα απαντήσουν. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίση θα ήθελα επειδή έχουμε ακόμα κάποιους συντονιστές στην αίθουσα και εσείς εκπροσωπείτε και τις διάφορες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, όλες, παρακαλώ προσπαθήστε να μιλήσετε με τους συντονιστές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Εμείς έχουμε αρκετά πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μια επίσκεψη στη συγκεκριμένη περιοχή της Ευρώπης θα μπορούσε να είναι μία ε, για να μπορέσουμε να δούμε μας τι συμβαίνει, ε, για να μπορέσουμε να δούμε ένα ακόμα ακαθόδε ζήτημα στην Ισπανία. Κάναμε μόλις μια αποστολή για άλλο θέμα για τα απαγωγέ παιδιών και αυτή είναι μια ακόμα πολύ παλιά ιστορία που πρέπει κάπως να επιληθεί. Υπάρχει κι άλλος τρόπος, αλλά προκειμένου να γίνουν όλα αυτά και να γίνει αποστολή πρέπει να υπάρξει και πλειοψηφία στην Επιτροπή μεταξύ των συντονιστών. Δεν ε, επαφείται σε μένα ή σε οποιονδήποτε άλλο, οι συντονιστέ αποφασίζουν και αυτό λοιπόν ε, είναι απλώ μια ε, προτροπή να αποτανθείτε στις πολιτικές σας ομάδες και να προσπαθήσετε να πιέσετε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Και όλες εσείς που ταξιδέψατε τόσο μακριά για να έρθετε στην καρδιά της Ευρώπης, της Βρυξέλλες, παρά το γεγονός ότι η καρδιά σας στην Ευρώπη είναι κάπου αλλού που είναι πολύ πιο ηλιόλουστα και πολύ πιο όμορφα για να είμαι ειλικρινής. Σας εύχομαι πραγματικά ε, καλή επιστροφή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δέσμευσή σας και γιατί διαβιβάσατε αυτές τις τόσο συγκινητικές ε, ιστορίες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουν απομείνει λίγοι συνάδελφοι στην αίθουσα. Ας καλωσορίσουμε τον επόμενο αναφέροντα. Πρόκειται για την αναφορά 760. Επίσης ισπανική αναφορά. Να ζητήσουμε από όσους εγκαταλείπουν την αίθουσα να κάνουν ησυχία. Και τον κύριο Χέσου Καρσόν ε, καλωσορίζω και τον παρακαλώ να πάρει το λόγο. Νομίζω ότι θα δούμε και μια παρουσίαση PowerPoint. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. να εκφράσουμε και εμείς την αλληλεγγύη μας και την υποστήριξή μας στην ομάδα για την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη που υποφέρει από την ε, νομική και δικαστική εγκατάλειψη που δεν κατάφεραν ακόμα να βρουν λύσεις σε όλα αυτά τα εγκλήματα να τους διαβεβαιώσουμε για την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη των περιβαλλοντικών ομάδων της Ισπανίας. Εδώ αντικαθιστώ έναν άλλο συνάδελφο, ο οποίος ε, έχασε τη ζωή του στην Αργεντινή πρόσφατα εργαζόμενος για την προστασία του περιβάλλοντος και είναι μεγάλη τιμή για μένα που τον αντικαθιστώ. Προφανώς το θέμα που έχουμε σήμερα είναι εντελώς διαφορετικό, αλλά έχει σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ο σεβασμός του περιβάλλοντος, ο σεβασμός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, της βιοπικιλότητας, της οδηγίας Habitat και επίσης ε, ο σεβασμός των διεθνών συμβάσεων για την βιοπικιλότητα, σύμβαση που έχει ε, επικυρωθεί από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα στην Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη είναι σημεία βιοπικιλότητας και φλεώδη για το περιβάλλον και παίζουν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο για την τροφιμική αλυσίδα και για την επιβίωση των ειδών. Υπάρχουν πολλά είδη λοιπόν άγριων πτηνών ιδιαίτερα τα οποία προστατεύονται στα πλαίσια της οδηγίας Habitat. Εδώ βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές τα φυσικά περιβάλλοντα στην Μεσόγειο έχουν υποστεί πάρα πολλές διαβρώσεις και ε, γενικά βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω ακριβώς ε, της ε, επιθυμίας των ανθρώπων, των κατοίκων της περιοχής ε, να τα εκμεταλλευτούν, να χτίσουν, να χρησιμοποιήσουν τα υλικά για κατασκευή σκαφών, σπιτιών κτλ. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που έχουν φυγεί ακόμα περισσότερο όπως η Τραμουντάνα, η αλυσίδα των ωραίων Τραμουντάνα όπου υπάρχει ε, ένα πρόγραμμα προστασίας του λεγόμενου μαύρο γήπα Υπάρχουν και άλλα είδη τα οποία είναι αντικείμενα προστασίας ε, στις Βαλεαρίδες νήσους από το 2008 υπάρχει ένας νόμος συμπληρωματικός της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που επέτρεψε σε ένα πληθυσμό ο οποίος ήταν ε, ε, σχεδόν εξαφανισμένος με βάση την διεθνή συνεργασία να ανακάμψει να περάσει από ε, μηδέν ζεύγια αναπαραγωγή σε 40 πλέον τέτοιου είδους ζεύγια. Εδώ βλέπετε το βόρειο τμήμα της νήσου Μαγιόρκα όπου συναντάμε τις ζώνες πλήρους προστασίας όπως επίσης και τις ειδικέ ζώνες εξαιρετικής, εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Τώρα όμως κάποιες από τις ζώνες αυτές απειλούνται από τον μαζικό τουρισμό και αγνοώντας τις διεθνείς συμβάσεις και τις εθνικές ρυθμίσεις η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων άνοιξε τις περιοχές αυτές σε τουριστικές δραστηριότητες. Και γι' αυτό θα δώσω τώρα τον λόγο στον συνάδελφό μου, ο οποίος είναι επιστήμων που ασχολείται με τα συγκεκριμένα θέματα. Είμαι από το Πανεπιστήμιο Αλκαλά και έχουμε κάνει μια μελέτη για τις ε, επιπτώσεις που θα έχει η αλλαγή του νόμου περιβαλλοντικής προστασίας που υιοθετήθηκε στις Βαλεαρίδες τον προηγούμενο χρόνο. Δύο είναι τα σημεία στα οποία θα σταθώ. Η οροσυρά Τραμουντάνα είναι κάτι το οποίο καλύπτει το 3 με 4% της ε, ε, νήσου και εκεί απαγορεύεται η είσοδος ε, των πολιτών εκτός όταν έχουν αδειοδοτηθεί για επιστημονικούς λόγους. Έτσι λοιπόν αυτές οι μικρές ζώνες οι οποίες είναι ζωτικές για τη διατήρηση της βιοπικιλότητας όχι μόνο της Μαγιόρκα αλλά και των Βαλεαρίδων να διατηρηθούν. Τώρα είναι σε κίνδυνο. Ε, ο τουρισμός είναι μαζικός. Εκατοντάδες χιλιάδες ε, άνθρωποι τώρα πια επισκέφτονται την οροσυρά της Τραμοντάνα. Και γι' αυτό έχουμε θέσει το θέμα και στις αρμόδιες ε, υπηρεσίες και στο Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος της Ισπανίας και την Περιφερειακή Κυβέρνηση και ο νόμος αυτός για την αλλαγή χρήσης είναι τεχνικού χαρακτήρα υποτίθεται, δεν υπάρχει όμως τίποτα που να το αποδεικνύει αυτό. Ακόμα και ο διαμεσολαβητής της Ισπανίας έθεσε ερωτήσεις στην κυβέρνηση των Βαλεαρίδων ε, για να μάθει ποια είναι τα τεχνικά αυτά στοιχεία, δεν πήρε καμία απάντηση έγινε μια διμερής συνάντηση για την αρμοδιότητα των περιοχών ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και την περιφερειακή κυβέρνηση αλλά δεν υπήρξε καμία αξιολόγηση των κινδύνων. Ε, η απόφαση λοιπόν αυτή όπως είπα ανοίγει όλα τα μονοπάτια και όλες τις εισόδους της περιοχής αυτής και αυτό θα προκαλέσει ουσιαστικά μια αλλαγή στη νομική ρύθμιση η οποία ίσχυε μέχρι τώρα και επιτρέπει την είσοδο περιηγητών στις περιοχές αυτές οι οποίες όπως είπα είναι ζώνες ζωτικής αναπαραγωγής ορισμένων ειδών και υπάρχουν προσπαθίες που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια ακόμα και με χρήματα και πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυστυχώ όμως ο τουρισμός ο μαζικός φτάνει στην οροσυρά της Τραμοντάνα και δεν αφήνεται λοιπόν κανένα μέρος, κανένα χώρος της νήσου στον οποίο να μην υπάρχει ελεύθερη είσοδος για τον τουρισμό και δεν υπάρχει καμία τεχνική τεχνηρίωση η οποία να λέγει ότι θα μπορούσε να γίνει και να επιτραπεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο κύριος Σιπριάνη και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η αναφορά έχει να κάνει με τις νέες διατάξεις που υιοθέτησαν οι περιφερειακές αρχές των Βαλαιαρίδων νήσων. Έχουμε εξετάσει αυτές τις διατάξεις και έχουν να κάνουν με τον ε, προγραμματισμό και την αδειοδότηση δραστηριοτήτων εντός των προστατευμένων περιοχών. Επιτρέπουν πιθανές χρήσεις όπως είναι η ε, δημόσια πρόσβαση, η διέλευση εντός αυτών ε, των αποκλεισμένων και προστατευμένων περιοχών. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης της περιοχής ε, ή σύμφωνα με ειδική αδειοδότηση και εξαρτάται από υποχρεωτική έκθεση των ε, αρμοδίων αρχών ε, που επιβεβαιώνει την συμμόρφωση με τον στόχο διατήρησης των τόπων αυτών. Εξετάσαμε την τεκμηρίωση που μας έστειλε στις 4 Οκτωβρίου αναφέρον, πριν λίγες μέρες δηλαδή. και γνωρίζουμε επίσης ότι έχει πραγματοποιηθεί διαπραγμάτευση ανάμεσα στις περιφερειακές αρχές των Βαλεαρίδων, νήσων και την κεντρική κυβέρνηση στη Μαδρίτη σχετικά με αυτές τις διατάξεις. Οι διαπραγματεύσεις αυτές στόχο είχαν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των νέων ε, διατάξεων με την Ισπανική νομοθεσία. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών ε, επιτεύχθη τον Ιούνιο, πριν λίγους μήνες δηλαδή, με συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις αυτές θα εφαρμόζονται με πλήρη συμμόρφωση του Ισπανικού Εθνικού Δικαίου για την εθνική κληρονομιά και την βιοπικιλότητα. Νομοθεσία που μεταφέρει και, εφαρμόζει την ε, οδηγία του βιότοπους ε, στην Ισπανία. Η συμφωνία αυτή σημαίνει ότι οποιαδήποτε απόφαση περιορισμός, ε, απαγόρευση δραστηριοτήτων στις προστατευμένες περιοχές ε, θα ρυθμίζεται εντός του σχεδίου διαχείρισης των τόπων αυτών ε, και θα βασίζεται στις ανάγκες των τόπων αυτών που σχετίζονται με τη διατήρηση των ειδών. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι οι διατάξεις αυτές ε, συμμορφώνονται με την εθνική ισπανική νομοθεσία. Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις πληροφορίες και κυρίως το γεγονός ότι οι νέε περιφερειακές διατάξεις στι Βαλεαρίδες νήσου θα ερμηνευτούν και θα εφαρμοστούν ε, σύμφωνα με το Ισπανικό Δίκαιο που ε, μεταφέρει στο Ισπανικό Δίκαιο τι οδηγίε για του βιότοπους και τα πτηνά. Θεωρούμε ότι δεν ε, υπάρχει ε, καμία παραβίαση των διατάξεων στις δύο αυτές οδηγίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ εσάς για μια πολύ σύντομη και σαφή απάντηση. Δεν είναι πάντα τόσο ε, στοχευμένες οι απαντήσεις. Δίνω το λόγο στους αδέρφους. Πρώτα η Ρώσα. Παρακαλώ. Ναι το επιθυμητό θα ήταν αυτό το οποίο ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή η νομοθεσία που εγκρίνει η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων να ε, μεταφέρει την νομοθεσία για το, η πολιτιστική κληρονομιά, διότι είναι αυτή η νομοθεσία που μετέφερε τη σχετική οδηγία και είναι η βασική νομοθεσία για την ε, περιβαλλοντική προστασία. Οι ε, αναφέροντες ήρθαν εδώ γιατί η προσαρμογή αυτή δεν γίνεται και αυτό που μας ανέφεραν οι αναφέροντες είναι ότι αυτή η τροποποίηση στην νομοθεσία ε, της ε, περιβαλλοντικής ε, αξιολόγησης και της εκτίμησης περιβαλλοντικών υποπτώσεων αντιβαίνει τη βασική νομοθεσία και επομένως και την οδηγία Habitat. Αυτό λοιπόν το οποίο θα ήθελα να ζητήσω είναι να παραμείνει ανοιχτή αναφορά, να δούμε με αποστολή επιστολών αν όντως αυτό ε, ε, θα το τηρήσουν και τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κλείσει η αναφορά. Αν όχι, να γίνουν όλες οι σχετικές έρευνες. Θα στείλουμε επιστολή στην κυβέρνηση και στην αντίστοιχη Κοινοβουλευτική Επιτροπή που συζητά τα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και ανάλογα με τις απαντήσεις που θα λάβουμε θα αποφασίσουμε. Δεν ξέρω εάν συμφωνούν οι αναφέροντες με αυτή τη δυνατότητα. Ναι, νομίζω εξαιρετική, διότι πράγματι η θεωρία που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ότι η αυτόνομη κυβέρνηση θα το λάβει υπόψη της, δεν είναι πολύ ωραία ημέρα βέβαια για να μιλάμε για τις αυτόνομες περιφέρειες στην Ισπανία σήμερα, αλλά αν όντω ε, γίνουν αυτά τα οποία είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς συμφωνούμε απολύτως ε, και ε, συμφωνούμε. Εμείς εκπροσωπούμε ένα πανεπιστήμιο και μια κυβερνητική οργάνωση. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον. Απλώς αυτές οι περιοχές οι οποίες ε, χρησιμοποιήθηκαν για την διατήρηση ενός πολύ σημαντικού είδους ε, ε, και γενικά των διαφόρων ειδών να παραμείνουν περιοχές Natura. Δεν ξέρω αν θέλει να πει ο συνάδελφος κάτι. Ναι, απλώς να προσθέσω ότι είναι πολύ ειδικέ οι περιστάσεις του συγκεκριμένου είδους αυτού του μαύρου γήπα. Βρίσκεται σε όλα τα νησιά της Μεσογείου και εξαφανίστηκαν και μόνο ένα μικρό μέρος τους ε, ζει στην Ισπανία και καταφέραμε να τα επανεισάγουμε στη Γαλλία και στι Βαλεαρίδες και το ιδιαίτερο αυτού του είδους είναι ότι αναπαράγεται πρακτικά όλο το χρόνο. Ε, τα Χριστούγεννα τον Ιανουάριο ήδη είναι στις φουλιές ε, και φέρνουν κλαδιά για να φτιάξουν, να χτίσουν τη φωλιά τους και μετά ε, γεννούν ένα μόνο αυγό. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ευαίσθητο είδος λοιπόν, το οποίο ε, αναπαράγεται σε δύο μήνες, ε, γεννιέται τον Απρίλιο ή τον Μάιο, είναι μια εποχή που ακόμα έχει πολύ κρύο στα βουνά και οποιαδήποτε ενόχληση, ακόμα και μισή ή μία ώρα να περάσει κάποιος από την περιοχή αυτή, τρομάζουν οι γονείς και φεύγουν από τη φωλιά και το ε, μπορεί ή το αυγό να σπάσει ή να φύγει και να πεθάνει από το κρύο το, ε, το μικρό, το νεογνώ. Πρέπει να το φροντίζουν, πρέπει να του δίνουν νερό επίσης να μην πεθάνει από τη δίψα αργότερα. Πρόκειται λοιπόν για μια αναπαραγωγική περίοδο η οποία ξεκινάει από 1η Ιανουαρίου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου διότι μετά από το πρώτο κρύο πρέπει να επιστρέψουν και πάλι στη φωλιά για να ξεκουραστούν και να ε, δυναμώνουν σιγά σιγά. Πρόκειται για ζώα που μπορούν να ζήσουν 50-60 χρόνια αλλά μέχρι τα 5-6 τους δεν αναπαράγονται. Που σημαίνει ότι οποιαδήποτε απώλεια μιας, ε, ε, ενός μικρού νεογνού σημαίνει ότι μπορεί να ε, επηρεάσει την αναπαραγωγή όλου αυτού του είδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν οι αναφέροντες νιώθουν εσά στο σπίτι τους και παίρνουν μόνοι τους το λόγο. Είναι σαν να τρώμε στο τραπέζι της κουζίνας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και Καλώ την κυρία Αλμπιόλ να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τους αναφέροντες για την παρουσία τους εδώ για το ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύουν για την προστασία του περιβάλλοντος ημεριζόμαστε την ανάγκη προστασίας του Μαυρογήπα Εγώ γνωρίζω περί ε, πρόκει, πρόκειται, προέρχομαι από την περιοχή της Βαλένθια, ξέρω τις αρνητικές συνέπειες που έχουν οι μαζικές ε, ε, κατασκευές, οικοδομές και τα λοιπά στο φυσικό περιβάλλον και σε ποιο βαθμό θέτουν σε κίνδυνο πάρα πολλά είδη. Γνωρίζω λοιπόν περί πρόκειται. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να τεθούν όρια σε συγκεκριμένες περιοχές για την προστασία τους. Το θέμα είναι ότι η κατάσταση εδώ έχει αρχίσει να, να στραβώνει γιατί υπάρχει μια οικογένεια η οποία είναι από τις πλουσιότερες στην Ισπανία και η οποία είναι ιδιοκτήτρια κάποιων εδαφών τα οποία ελέγχουν την είσοδο στις περιοχές αυτές. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες γι' αυτό και για τις οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος γιατί το θέμα είναι ότι η δεξιά στη Μαγιόρκα που είναι στην κυβέρνηση αφού ε, ε, κατέστρεψε το φυσικό περιβάλλον υποτίθεται ότι κόπτεται τώρα για την προστασία των μαυρογυπών. Κοιτάξτε, ε, δεν είναι θέμα για να συζητήσουμε εσωτερικά πολιτικά θέματα, παρακαλώ. Θα πρέπει να παραμείνετε στη συζήτηση των θεμάτων τα οποία έχουμε μπροστά μας και αν έχετε να κάνετε πολιτικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις να τις κάνετε εκτός εθούσης. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο ζητώ εγώ είναι όπως και όλες οι, όπως όλες οι παρεμβάσεις των βουλευτών που κάνουν αναφορές στις διάφορες κυβερνήσεις και εγώ μιλάω ε, για την κυβέρνηση ε, της, ε, των Βαλεαρίδων και να πω ότι έχει κάνει λάθη η κυβέρνηση λοιπόν των Βαλεαρίδων στην αλλαγή της χρήσης. Προφανώς θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τα λάθη αυτά και να ζητήσουμε να αποκατασταθούν έτσι ώστε να υπάρξει προστασία και να έχουμε όμως ανοιχτή την πρόσβαση στους, στο λαό σε κάποιες περιοχές, να μην στερούμε την πρόσβασή τους σε περιοχές όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Προφανώς και θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, το περιβάλλον και έχουμε και το παράδειγμα ε, της ε, περιοχής του Μορτής όπου επιτρέπεται είσοδος αλλά υπάρχουν περιορισμοί στην κίνηση μέσα στην συγκεκριμένη ζώνη. Εμείς λοιπόν θέλουμε να προστατευθεί η περιοχή αυτή, να υπάρξουν πάρα πολλές ε, φυσικά ε, να υπάρξουν πάρα πολλοί περιορισμοί την εποχή όπου υπάρχει η διαδικασία αναπαραγωγής και όλα αυτά τα μέτρα να ληφθούν επί τη βάση επιστημονικών μελετών. Αυτή είναι η θέση μας σε σχέση με τη συγκεκριμένη αναφορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ιστούρης Βουάιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα πέσω σε αυτό το πολιτικό τερτύπι που έκανε η συνάδελφος και θα ήθελα να το σημειώσει η Επιτροπή. Δυστυχώς ε, είναι σύνηθες αυτό το φαινόμενο. Ξέρουμε ποιος στηρίζει και ποιος δεν υποστηρίζει. Ε, εγώ μιλάω για την ε, Ισπανία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαμε να την παρατείνουμε αυτή η πολιτική συζήτηση, αλλά όπως είπε η Πρόεδρος, δεν είναι ούτε η στιγμή, ούτε ο χώρος να γίνει αυτή η συζήτηση. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια της κυρίας Αλβιόλ. Να σημειώσει η Πρόεδρος ότι με διακόπτει συνεχώς. Αυτό είναι ο δημοκρατικός χαρακτήρας της συντρόφου, το γνωρίζουμε δυστυχώς. Ε, εδώ και τρία χρόνια το γνωρίζουμε το χαρακτήρα στο Κοινοβούλιο. Εγώ δεν μίλησα. Οι παρεμβάσεις δυστυχώς που γίνονται προς τη μία προς την άλλη κατεύθυνση πρέπει να ακούγονται. Πρέπει να ακούμε και τα θετικά και τις επικρίσεις. Να τα αναλύουμε και να δούμε ότι σε αυτή την περίπτωση πράγματι ε, αναφερόμαστε σε μία υπόθεση που αφορά το περιβάλλον τις ε, Βαλαρίδες και πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση των Βαλαρίδων όπως και σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση να δραστηριοποιηθεί και να κάνει την πορεία για την υπόθεση αυτή. Ε, είναι αρκετοί οι λόγοι, η προστασία του περιβάλλοντος κυρίως, ε, υπάρχει νομοθεσία ισπανική η οποία δεν τηρείται και εγώ θα έκανα μία έκκληση όχι σε πολιτικό επίπεδο, το αντίθετο, να ε, επιστρέψουμε στην νομιμότητα και να μην ε, ε, προκαλούμε ανασφάλεια όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς σε διάφορες περιοχές στην Ισπανία κοντά στη Μεσόγειο γίνονται αλλαγές στην νομοθεσία οι οποίες προκαλούν έλλειψη ασφάλειας δικαίου όπως γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ε, να επικεντρωθούμε σε αυτό μόνο και να ακούσουμε γιατί, ε, τους εμπειρογνώμονες, γιατί γι' αυτό υπάρχει επιτροπή, ε, διότι υπάρχει παραβίαση του νόμου από την κυβέρνηση των Βελαρίδων, υπάρχει χρόνος να επανορθώσει και φυσικά με την εποπτεία και τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ένα διαδικαστικό δεν απαγορεύεται πουθενά στην κοινωνία ούτε στην πολιτική ε, μεταξύ ευρωβουλευτών να χρησιμοποιούν ευγένεια, κοινή λογική και λίγη κομψότητα. Αυτό απαιτείται και είναι χρήσιμο να εφαρμόζεται από όλους. αλλού θα πρέπει να διεξάγονται οι πολιτικές μάχες, όχι στην αίθουσα της Επιτροπής μου. Κλείνοντας με αυτήν τη θετική παρατήρηση, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε από τόσο μακριά και που μας μεταφέρατε το μήνυμά σας, τα επιστημονικά σας στοιχεία. Ε, λάβαμε γνώση και θα ήθελα να συνοψίσω. Θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει γραπτό τις πληροφορίες που μας έδωσε. Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να στείλουμε επιστολή στις αρχές των Βαλεαρίδων νήσων, να αναφέρουμε ε, ότι μας επισκέφθηκαν οι εμπειρογνώμονες ε, και η επιστολή αυτή θα σταλεί και στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ισπανίας εδώ στις Βρυξέλλες, ε, ενημερωτικά λέγοντάς τους ότι παρακολουθούμε το θέμα αυτό, διότι η πλήρης συμμόρφωση με την οδηγία ε, είναι θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή μας. Θέλουμε λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι δεν θα υπάρχουν δυσκολίες ως προς αυτό το θέμα. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο συνάδελφο το λόγο. Μπορείτε να συμφωνήσετε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή επιστροφή ε, στην όμορφη Μαγιόρκα. Με τις καλύτερες ευχές μας. Ελπίζουμε σύντομα να επισκεφτούμε και εμείς ε, τη Μαγιόρκα σύντομα. Κάποια στιγμή. Το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η αναφορά 1304. Άλλη μια ισπανική αναφορά, διαφορετικό θέμα όμως έχει να κάνει με τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας των πανεπιστημιακών διδασκόντων ορισμένου χρόνου. Νομίζω ότι είναι παρόντες οι αναφέροντες. Καλωσορίζω την Ισαβέλ Τελακρούς και τον Μινθέντ Μονρόικ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πέντε λεπτά συνολικά να τα μοιραστείτε μεταξύ σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ σήμερα για να σας εξηγήσουμε την αναφορά την οποία σας έχουμε καταθέσει για τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες μιας μεγάλης ομάδας οργανωμένων ε, καθηγητών ανδρών και γυναικών του Πανεπιστημίου της Βαλένσια ε, που είναι αναγνωρίζεται ως βοηθητικό προσωπικό και ερευνητικό προσωπικό. Έχουμε προσπαθήσει να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα με πάρα πολλές συναντήσεις με τις πανεπιστημιακές αρχές, με τον ε, με τον Κοσμήτορα, με την υπεύθυνη του καθηγητικού σώματος, με την περιφερειακή κυβέρνηση, με τη Γενική Διεύθυνση των Πανεπιστημίων, με όλες τις πολιτικές ομάδες οι οποίες συναποτελούν ε, το Κοινοβούλιο της Βαλένθια. Δυστυχώς αποτύχαμε η επισφαλής κατάσταση, οι διακρίσεις τις οποίες υφιστάμεθα σε επίπεδο συνθήκων εργασίας και σε επίπεδο αμοιβών δεν χαρακτηρίζει μόνο το Πανεπιστήμιο της Βαλένσια αλλά όλα τα δημόσια πανεπιστήμια. Στο Πανεπιστήμιο της Βαλένσια στη δική μας περίπτωση οι άνδρες και γυναίκες που εργάζονται εκεί που έχουμε περάσει φυσικά στο Πανεπιστήμιο μετά από ειδικέ εξετάσεις αντιπροσωπεύουμε το 1 τρίτο του καθηγητικού προσωπικού. Υπήρχαν το 2016 1.246 καθηγητές ε, τέτοιου, ε, αυτής της κατηγορίας. Ε, νομίζω ότι αντιπροσωπεύουμε ουσιαστικά το 41% όλων των θέσεων του Πανεπιστημίου, των θέσεων εργασίας του Πανεπιστημίου μας, σε επίπεδο καθηγητικού προσωπικού. Αντιπροσωπεύουμε 13,5 credits ε, και ουσιαστικά αντιπροσωπεύομαι θα έλεγα συνολικά σε όλα τα επίπεδα και ε, τις βαθμίδες το 75% των διδασκόντων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν ο ρόλος μας για την σωστή λειτουργία του Πανεπιστημίου και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να υφιστάμεθα αυτές τις διακρίσεις. Καταρχάς, οι μισθολογικές συνθήκες του προσωπικού αυτού είναι πραγματικά ακατάλληλες σε επίπεδο των απαιτούμενων προσόντων και είναι πάρα πολύ χαμηλότερα σε σχέση με άλλες κατηγορίες διδασκόντων. Για να καταλάβετε, ένας κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου, ένας καθηγητής, όχι ένας δόκτωρ, μπορεί να φτάνει σε 6.213 ευρώ. Ε, ένας καθηγητής μπορεί να φτάνει και τις 7.000. Είναι σαφές ότι ήδη εδώ έχουμε μία διάκριση σε σχέση ε, με τις αμοιβέ. Αν δούμε πραγματικά πόσες ώρες εργάζεται κάποιος, σύμφωνα με τα έγγραφα που δίνει το ίδιο το Πανεπιστήμιο, για κάθε ώρα εργασίας χρειάζονται 7 ώρες για την προετοιμασία, ε, για συνάντηση με τους ε, φοιτητές, για συνεργασία με το υπόλοιπο καθηγητικό προσωπικό κτλ. Και υπάρχει προσωπικό που εργάζεται μόνο δυστυχώς βοηθητικό με 5,13 ευρώ την ώρα. Αυτό το 5,43 συγγνώμη ε, την ώρα είναι καταλαβαίνετε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που ζήσαμε πρόσφατα. Το 2012 ήμασταν πολύ λιγότεροι, τώρα υπάρχει μία αύξηση, έχουμε φτάσει τους 1246, είναι δεδομένα επίσημα αυτά, ήμασταν 974 και δεύτερον το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τέτοιου είδους συμβάσεις τις οποίες ανανεώνει σε ετήσια, εξαμηνιαία ή τριμηνιαία βάση και δημιουργείται μια συνεχής αντικατάσταση του προσωπικού η οποία μπορεί να γίνεται πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας ενός ε, διδάσκοντος. Έτσι λοιπόν, ε, ε, αυτές οι επαγγελματικές, οι εργασιακές μάλλον πρακτικές δεν θα επιτρέπεται να, θα να γίνουν σε καμία επιχείρηση σύμφωνα με τους κανόνους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνθήκες εργασίας, σε πάση περιπτώσει, είναι απαράδεκτες τα εργασιακά δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται στις επιχειρήσεις τις μεμονωμένες δεν αναγνωρίζονται στην περίπτωση αυτή. Το Πανεπιστήμιο της Βαλένσια δεν αναγνωρίζει όπως άλλα ιδρύματα ε, την εργασιακή ε, νομοθεσία. και μάλιστα μειώνονται και οι ώρες απασχόλησης σε όλες τις κατηγορίες των καθηγητών εκτός από τις δικές μας. Όπως φαίνεται από τα τελευταία έγγραφα βλέπουμε ότι το κέρδος από τη μείωση των ωρών του ωραρίου εργασίας είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να χαρακτηρίζει ε, την δική μας επαγγελματική κατηγορία. Υπάρχει λοιπόν μια διάκριση και σε επίπεδο ωραρίου εις βάρος της δικής μας κατηγορίας. και δεν μπορούμε εμείς έτσι με τον τρόπο που εργαζόμαστε να συμμετέχουμε σε ανταγωνιστικές διερευνητικές ομάδες. Αυτό δείχνει για μια ακόμη φορά τις διακρίσεις τις οποίες υφιστάμεθα και το ίδιο συμβαίνει και με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται οι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο, η δική μας τουλάχιστον κατηγορία, ακόμα και αν έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 12 ετή για να μπορέσουν να διεκδικήσουν ορισμένες θέσεις. Ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλές επίσης δυνατότητες προαγωγής αν θέλετε ε, σε διάφορες κατηγορίες του επιστημονικού προσωπικού εκτός από την δική μας κατηγορία. Δεν γίνονται λοιπόν σεβαστά τα δικαιώματά μας και κάθε χρόνο οι συνθήκες αυτές ε, ανανεώνονται για μια ακόμη φορά ε, και λειτουργούμε σε ετήσια βάση ακόμα και αν δουλεύουμε 25 ολόκληρα χρόνια και παραμένουμε ουσιαστικά εκτός δυνατότητας επιρροής της οργάνωσης η οποία μας ε, απασχολεί, είναι ο εργοδότης μας. Υπάρχει λοιπόν με ένας αποκλεισμός και μία μορφή εκμετάλλευσης του προσωπικού καταγγέλουμε την εκμετάλλευση αυτή. Θα πρέπει να ζητήσουμε και να ζητήσετε την καταγγελία αυτής της απαράδεκτης κατάστασης όχι για τη δική μας αν θέλετε βελτίωση αλλά για την βελτίωση των ίδιων των πανεπιστημίων στα οποία απασχολούμεθα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τη δική της άποψη η κυρία Ποκόρνη έχει το λόγο. Ο κύριος Ποκόρνη, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, αναφέροντες για την ε, ε, πλήρη παρουσίασή τους. Η προστασία της επισφαλούς απασχόλησης είναι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι τμήμα του κοινωνικού πυλώνα της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επίσης ιδιαίτερα η εφαρμογή της οδηγίας 70 του 1999 που ε, προστατεύει τους εργαζομένους με συνθήκες, με συμβάσεις ε, ορισμένου χρόνου. Υπάρχουν δύο παρατηρήσεις που πρέπει να γίνουν εδώ. Η οδηγία βασίζεται βασικά σε συμφωνία ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους. Η ρήτρα 4 προβλέπει τη συγκεκριμένη συμφωνίας ότι αυτοί οι οποίοι εργάζονται με ε, συμβάσει ορισμένου χρόνου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με ε, διακρίσεις σε σχέση με αυτούς οι οποίοι εργάζονται με συνθήκες ή κάτω από συνθήκες αορίστου χρόνου. Ο εισηγητής ο αναφέρον είπε ότι αυτή η κατάσταση επικρατεί εδώ και 25 χρόνια. Όπως είπα, εκτός και αν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι οι οποίοι οδηγούν στην επαναληπτικότητα της θέσης σε ισχύ αυτών των συμβάσεων και εκτός αν ο αριθμός των δυνατοτήτων του αριθμού αυτών που μπορούν να εργαστούν με τις συμβάσεις αυτές μειωθεί βλέπουμε ότι η σύγκριση ανάμεσα στους μονίμους και ε, στους απασχολούμενους με ορισμένο χρόνο ε, οι συνθήκες είναι μερικές φορές ε, πολύ χειρότερες για τους ορισμένου χρόνου από ό,τι για τους αορίστου. Η προστασία στα πλαίσια της οδηγίας αναφέρεται βέβαια κυρίως στα εργασιακά και στις συνθήκες εργασίας, αλλά τα παραδείγματα τα οποία μας δώσατε θα έλεγα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Έχουν σχέση επίσης και με τη γονική άδεια, την ετήσια άδεια, την άδεια για λόγους ασθενείας κτλ. Μας φαίνεται λοιπόν εμάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν ε, αποδείξεις εδώ για διακρίσεις ανάμεσα στις δύο κατηγορίες των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο της Βαλένσια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι η ρήτρα υπαριθμών 4 για την πρόληψη των διακρίσεων μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας, οπότε κανονικά οι αναφέροντες θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τους εθνικούς μηχανισμούς, ακόμα επίσης και την διαιτησία, για να ζητηθεί άμεσα η εφαρμογή της ρήτρας 4 της συγκεκριμένης οδηγίας. Σε σχέση τώρα με την διάρκεια, τη χρονική των παρατάσεων ή ανανεώσεων των συμβάσεων, είναι σαφές ότι η νομολογία μέχρι τώρα ήταν σαφεστάτη ότι οι παρατάσεις αυτές δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη μονίμων αναγκών. Δηλαδή οι έκτακτες συμβάσεις καλύπτουν έκτακτες ανάγκες. Αυτό είναι κάτι το οποίο τέθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2013, βγήκε απόφαση το 2014 και το δικαστήριο είπε, απεφάνθη ότι η εθνική νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται στην Ισπανία δεν παραβιάζει την συγκεκριμένη ρήτρα της οδηγίας. Παρόλα αυτά αναφέρθηκε επίσης και στα εθνικά δικαστήρια και ζήτησε τα εθνικά δικαστήρια να κρίνουν αν σε ένα πανεπιστήμιο της Καταλωνίας οι συνθήκες ήταν αντίστοιχες με αυτές οι οποίες παρουσιάστηκαν από τους αναφέροντες. Το θέμα έχει περάσει τώρα στο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο είπε ότι οι συμβάσεις ήταν άκυρες γιατί δεν είχαν γίνει σεβαστές οι ρυθμίσεις τις οποίες προβλέπει η εθνική ισπανική νομοθεσία. Η άποψή μας είναι ότι η απόφαση αυτή δίδει μια ερμηνεία του εθνικού δικαίου η οποία θα μπορούσε να ισχύσει και για το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια και είναι ένας ένομος τρόπος να ζητηθεί αποκατάσταση και αποζημίωση γιατί οι ρυθμίσεις λειτουργίας του Πανεπιστημίου δεν είναι συμβατές με τις ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. Το θέμα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο δημόσιο στην Ισπανία είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει στο παρελθόν και νομίζω ότι θα έχουμε ξανά την δυνατότητα να το συζητήσουμε μαζί σας σε μια μελλοντική ευκαιρία όταν προχωρήσουν οι συζητήσεις και όταν έχουμε διερευνήσει ακόμα περισσότερο την υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο σε συναδέλφους. Η κυρία Στανόκα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε το νομικό πλαίσιο και ευχαριστώ τους αναφέροντες που ήρθαν εδώ στην Επιτροπή μας. Έχουμε σαφή περίπτωση διάκρισης εφόσον μιλάμε για άνηση αμοιβή ε, για την ίδια δουλειά. Εγώ επί χρόνια ήμουν λέκτορα σε πανεπιστήμιο ε, στη Ρήγα. Ε, είναι πρόβλημα λοιπόν που αφορά συναδέρφους μου. Επίσης είμαι μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Και λέμε συνέχεια ότι αυτές οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν μπορούν να αποτελούν λύση σε μια σειρά προβλημάτων. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, επισφαλείς συνθήκες εργασίας, ε, τη μείωση των ε, αμοιβών σε όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μου και της Ισπανίας. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την οδηγία και την προφανή παραβίασή της. Αναφέρομαι στην οδηγία του 1999 Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, να στείλουμε επιστολή στις ε, αρμόδιες ε, ισπανικές αρχές όπου να περιγράφουμε τις ανησυχίες μας και να στείλουμε την αναφορά αυτή και ε, στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινών Υποθέσεων προς ενημέρωσή της. Έχουμε άλλωστε αρκετέ αναφορές ε, σχετικά με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Αλβιόλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η επισφάλεια στην απασχόληση είναι ένα δράμα το οποίο βιώνουμε στο Ισπανικό κράτος. Υπάρχουν πάρα πολλές συμβάσεις ορισμένου χρόνου με πολύ λιγότερα δικαιώματα από ότι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Είναι μια πολύ άσχημη πραγματικότητα η οποία δυστυχώς χαρακτηρίζει και τα δημόσια πανεπιστήμια και την δημόσια επίσης τις δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες χρησιμοποιούν εκπαιδευμένους σωστά, καταρτισμένους σωστά εργαζομένους με ελάχιστες αμοιβέ. Το 41% των πανεπιστημιακών θέσεων στην Ισπανία δυστυχώς είναι προσωρινές θέσεις απασχόλησης, είναι επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, αυτό είναι ένα δράμα για τους εργαζομένους, αλλά είναι ένα δράμα και για την ίδια την δομή των πανεπιστημίων και ιδιαίτερα των δημόσιων πανεπιστημίων. Οι συμβάσεις λοιπόν αυτές ορισμένου χρόνου ορίζονται φυσικά από ρυθμίσεις ε, για τις οποίες αποφασίζει η κάθε φορά το, το κράτος, το δημόσιο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση παίζουν ρόλο και οι ε, τοπικές κυβερνήσεις και περιφερειακές διοικήσεις. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια οδηγία Ευρωπαϊκή η οποία προβλέπει ότι οι συνθήκες εργασίας αυτών που έχουν ορισμένου χρόνου συμβάσει, δεν μπορεί να είναι χειρότερες από αυτούς οι οποίοι εργάζονται που είναι μόνιμοι ή που εργάζονται με συνθήκες αορίστου χρόνου. Οι επαφές με τις τοπικές αρχές έχουν ήδη γίνει όμως, δεν έχει υπάρξει μια λύση και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι όλα αυτά μπορεί να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο ε, νομικό στην Ισπανία, οι προσπάθειες έχουν γίνει, δεν, ήταν, ε, δεν ευωδόθησαν. Παραμένει λοιπόν το θέμα, είναι θέμα δικαιοσύνης, πρέπει να εξαντληθούν όμως όλοι, όλα τα νομικά μέσα τα οποία μπορεί να υπάρξουν αλλά νομίζω ότι και εμείς μπορούμε εμείς να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά ζητώντας από τις αρχές να πράξουν τα δέοντα. Να βάλω μία παρένθεση εδώ. Το θέμα αυτό είναι πολιτικό. Τι εννοώ με αυτό. Ε, και γιατί είμαστε κοινοβούλιο, αλλά γιατί η επισφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία των θυμάτων, είναι καρπός των αποφάσεων που λαμβάνουν ή δεν λαμβάνουν οι κυβερνήσεις μας. Επιμένω λοιπόν, όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα είναι βαθιά πολιτικά θέματα. Οι συνθήκες εργασίας είναι πολιτικό θέμα. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πολιτικό θέμα. Και δεν μπορούμε να μην τα αντιμετωπίσουμε με πολιτικό βλέμμα. αυτό κάνουμε εδώ, πολιτική και διάλογο δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά το να το κάνουμε με ευγενικό τρόπο είναι, θα έλεγα, κάτι το οποίο δείχνει την αξιοπρέπεια του ομιλούντος. Ο κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί αναφέροντες, από την περιγραφή της κατάστασης διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει αναλυτικά αυτήν την αναφορά. Και με βάση την ε, αναφορά και τις διατάξεις ε, του δικαστηρίου Οι διατάξεις αυτές αποτελούν πια εθνικό δίκαιο. Μπορείτε λοιπόν να προσφύγετε στα δικαστήρια της χώρας σας. Δέχομαι όμως και και το πάθος της κυρίας Γκούτσμαν μας δείχνει ακριβώς αυτό, ότι δεν είναι πάντα αξιόπιστη η κυβέρνηση όσον αφορά την εφαρμογή του εθνικού δικαίου, ούτε όταν μιλάμε για το ε, ευρωπαϊκό δίκαιο. Η επιρροή λοιπόν που μπορούμε εμείς να ασκήσουμε αυτή η ήπια εξουσία του της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στην ε, περίπτωση αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να περιμένουμε την ε, σχετική θέση της Επιτροπής Απασχόλησης, ε, διότι μπορεί και εκείνη να μπορεί να συνεισφέρει στο θέμα. Νομίζω όμως ότι και όσον αφορά τις διατάξεις ε, απασχόλησης και όσον αφορά το θέμα της αμοιβή, ε, μιλάμε για διακρίσεις. Θα πρέπει λοιπόν σε ένα πολιτισμένο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρείτε το δίκιο σας. Εμείς ε, λοιπόν θα απαιτήσουμε την εφαρμογή του δικαίου αυτού. Και γι' αυτό συμφωνώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή μέχρι η Επιτροπή Απασχόλησης ε, να μας ε, έχει υποβάλει την δήλωσή της για να μπορέσουμε να οργανώσουμε εκεί τον τρόπο που θα σας υποστηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριάς. Από τη συζήτηση προκύπτει ότι και στην Ισπανία συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Διότι και στην Ελλάδα έχουμε ένα σύστημα του Προεδρικού Διατάγματος 407. Διδάσκοντες του 407 λέγονται. Και είναι ε, επιστήμονες οι οποίοι προσλαμβάνονται για τρία χρόνια αλλά βέβαια δεν έχουν τις ίδιες αμοιβέ με όσους κάνουν την ίδια εργασία στο Πανεπιστήμιο. Και φυσικά παραβιάζεται η οδηγία του 1999, η οποία όπως και στην περίπτωση αυτή αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου χρόνου. Και πολύ περισσότερο, θα πρέπει να το δουν αυτό οι φίλοι από την Ισπανία, δεν θέλω να τους κάνω υποδείξεις, αλλά εάν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, τότε με βάση την οδηγία έχουν δικαίωμα να μετατρέψουν τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Και αυτό είναι επίσης κάτι σημαντικό. Ε, εγώ χρόνια είμαι πανεπιστημιακός και αντιμετωπίζαμε αυτό το ζήτημα στην Ελλάδα και θεωρώ ότι φυσικά πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία για να δώσει το δικαίωμα να μετατραπούν σε συμβάσει αορίστου χρόνου και όσων είναι με το Προεδρικό Διάταγμα 407 και φυσικά και στην περίπτωση των συναδέλφων από την Ισπανία. Το δεύτερο που έχει σημασία έχει σχέση και δεν το άκουσα, ίσως μέχρι να έρθω παρακολουθούσα από το monitor τη συζήτηση, αλλά στο διάστημα μέχρι να έρθω μπορεί να υπόθηκε. Υπάρχει μία επίπτωση και στο συνταξιοδοτικό, διότι εφόσον παίρνουν λιγότερα χρήματα από εκεί και πέρα και η σύνταξή τους είναι σε διαφορετικό επίπεδο. Άρα λοιπόν η διάκριση δεν αφορά μόνο τα ποσά που παίρνουν σήμερα, τις συνθήκες με τις οποίες απασχολούνται σήμερα, αλλά και το χρόνο στον οποίο θα βγουν σε σύνταξη, καθώς επίσης και το ποσό με το οποίο θα βγουν στη σύνταξη. Επομένως εδώ, όπως υπόθηκε και από άλλους συναδέλφους, έχουμε παραβίαση της οδηγίας του 1999. Προφανώς μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στα δικαστήρια της Ισπανίας για να υπάρξει μια διαδικασία όπου θα αναγκαστεί η κυβέρνηση να τηρήσει την νομοθεσία. Βεβαίως η Κομισιόν έχει αφήσει ανοιχτό το ζήτημα αν ε, συνεχίζει να είναι αυτό μια πρακτική της Ισπανίας κατά πόσο Βεβαίω θα μπορούσε να παραπεμφθεί και για παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, να έχουμε και την άποψη των συναδέλφων της Επιτροπής Απασχόλησης, αλλά βεβαίως όλα αυτά είναι όπως υπόθηκε πολιτικές επιλογές. Πολιτικές επιλογές της ευελιξίας, πολιτικές επιλογές να έχουμε άλλους εργαζόμενους με ε, περιορισμένου χρόνου συμβάσει άλλου με αορίστου, διότι το σύστημα το ίδιο δεν επιθυμεί να ομαλοποιήσει όλες τις διαδικασίες. Και πολύ περισσότερο στα πανεπιστήμια, όπου εκεί πρέπει να τηρείται ο νόμο, Μια και στα πανεπιστήμια και στις νομικές σχολές διδάσκουμε την τήρηση του νόμου. Ευχαριστώ πολύ. Thank ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θυμίσω στους συναδέλφους ότι σήμερα το πρωί μεταξύ των συντονιστών είχαμε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την ε, ακρόση που θα οργανώσουμε στις 22 Νοεμβρίου που ε, έχει τον τίτλο «Προστασία των εργαζομένων σε επισφαλείς ε, συνθήκες εργασίες και στην προσωρινή εργασία» ακρόαση αυτή θα μεταδοθεί από το διαδίκτυο. Μπορείτε λοιπόν να την παρακολουθήσετε από τη Βαλένθια. Θα διαρκέσει κάποιες ώρες και θα ε, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα όπου θα συμμετάσχουν διάφορες ομάδες συμφερόντων. Ε, συνήθως ε, μάλιστα οι ε, μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι η McDonald's ε, εκμεταλλεύεται ε, τους εργαζομένους. Τώρα όμως μιλάμε για πανεπιστήμια. Βλέπουμε λοιπόν ε, πολύ ευρύ πεδίο όπου βλέπουμε το φαινόμενο αυτό. Είναι λοιπόν ε, κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δεν μας παίρνει να έχουμε οργανικές διαμάχες ε, το θέμα αυτό. Θα πρέπει να βρισκόμαστε στο πλευρό των Ευρωπαίων πολιτών και να αποτελεί προτεραιότητα για μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή, να την ε, στείλουμε επίσης στην Επιτροπή Απασχόλησης προ ενημέρωσή της και ε, παραθέτω και τα λόγια του εκπροσώπου της Επιτροπής ε, ότι βλέπουμε εδώ να υφίστανται διακρίσεις. Σας καλώ να απευθυνθείτε και στα, να προσφύγετε στα δικαστήρια της χώρας σας, διότι η άμεση οδός είναι ε, να προσφύγετε στα εθνικά δικαστήρια. Θα ε, συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση και μετά την πραγματοποίηση της ακρόασής μας και θα δούμε αν θα, μήπως ε, καταφέρουμε να έχουμε εκτενέστερο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω στο θέμα αυτό. Συμφωνείτε να προχωρήσουμε έτσι? Ωραία. Θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις. Διότι δεν είναι πολύ απλή υπόθεση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ξανακαλέσω να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ε, καταρχάς να ευχαριστήσουμε πολύ την ε, Επιτροπή για την δεκτικότητα και κιόλας που εμφανίζουν για ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για σημαντικό αριθμό εργαζομένων αλλά και για τους φοιτητές μας που είναι και το μέλλον μας διότι αυτό το οποίο βλέπουν, αυτό το οποίο αντιλαμβάνονται, αυτό το οποίο τους διαβιβάζουμε ε, μπορώ να πω ότι δεν είναι και το πλέον θετικό. Όσον αφορά την δικαστική οδό, προσφύγαμε στο δικαστήριο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά μόνο η δικαστική οδός δεν πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα, διότι μπορούμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο μόνο εκ των υστέρων και όταν έχει κάτι συμβεί, όταν δεν σου ανανεώνουν τη σύμβαση, όταν δεν σου δίνουν θέση εργασίας. Και αυτή είναι μια κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλοί άνθρωποι και ε, νομίζω ότι είναι ε, ε, μία απόφαση που πρέπει να τη λάβει η κυβέρνησή μας. Η αυτόνομη εθνική κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιος είναι ο αρμόδιος, αλλά θα πρέπει εσείς είπατε ότι θα πρέπει να τους διαβάσετε μια ανακοίνωση, μια επιστολή, δεν ξέρω εγώ τα ορολογία, τα ξέρετε εσείς και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν είναι πάντα η δικαστική οδός αυτή η οποία μας ενδιαφέρει. Ε, μας χρειάζεται αλλά όχι για όλους ε, ε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και μάλιστα υποφέρουμε πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτή την αλλαγή θα συνεχίσουμε λοιπόν να εξετάζουμε το θέμα, αλλά όπως είπατε και εσείς, είναι συστηματική η κατάσταση, δεν είναι πλέον ε, προσωπική και πραγματικά και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η αυτόνομη περιφέρεια της Βαλένθια θα λάβει τις πληροφορίες. Θα το παρακολουθούμε εμείς, αλλά όπως είπε και ο κύριος Μαριάς, ε, είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Επομένως, ε, είναι συστηματικού χαρακτήρα πλέον και ε, αυτό αποτελεί ένα μεν παράδειγμα, αλλά το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Αφορά τα πανεπιστημίνη της Ουψάλας, ε, της Αθήνας κλπ. Ε, επομένως ε, πρέπει πάντα να το εξετάζουμε. Και ξέρω ότι έχουμε και τους εκπροσώπους ε, του γραφείου της Βαλένθια εδώ σήμερα και είμαι βέβαιος, βέβαιη ότι το έχετε σημειώσει και το, θα τα αναφέρετε στις περιφερειακές αρχές όλα αυτά. Να προχωρήσουμε λοιπόν. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και ευχαριστώ και σε όλους εκείνους που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Περνάμε τώρα στην επόμενη αναφορά που είναι και αυτή η Ισπανική. Καλύπτουμε όμως ένα πολύ ευρύ φάσμα πολύ διαφορετικών αναφορών ε, από την Ισπανία σήμερα. Τώρα έχουμε την 161 για τις ε, πρακτικές της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Λογικά πρέπει να έχουμε εδώ και τους αναφέροντες, Σουζάνα Φερνάντες και Αλμπέρτο Αράν Σανταντέρ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Επιτρέψτε μου ε, καταρχάς να πω ότι είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να βλέπω Προεδρείο γεμάτο γυναίκες. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που μας επέτρεψαν να παρουσιάσουμε αυτή την πρόταση στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη Γραμματεία μέχρι και τους ευρωβουλευτές που βοήθησαν να φτάσουμε στην αναφορά μας. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε όλους εκείνους που δίνουν μάχη μαζί με μας ε, για την Ισπανική Εθνική Νομοθεσία, η οποία ε, ε, δεν λαμβάνει υπόψη στις οδηγίες που έρχονται του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να αναφέρω επίσης την Ειδική Ένωση Υποθηκών και μια πολύ καλή υπόμνηση στο άτομο το οποίο μας έδωσε πληροφορίες ε, για τις υποθήκες, το Χωσέ Μανουέλ Νοβόας. Έχουμε διάφορες ε, οργανώσεις ε, στην Καστήλη Λεών και πάρα πολλές οργανώσεις οι οποίες μας ακολουθούν σε αυτή τη μάχη καταγγέλουμε την άδικη κατάσταση την οποία βιώνουμε οι Ισπανοί καταναλωτές, αντίθετα με όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Η κυβέρνησή μας μεταφέρει τις οδηγίες που ε, τους βολεύουν για να εφαρμόσουν την πολιτική λιτότητα, ενώ όσον αφορά το ε, ε, σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών ε, δεν σέβεται καθόλου. Και αυτό έχουμε φτάσει στο σημείο να πρέπει να επιβάλλει κυρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας γιατί δεν τηρούν τις κατάλληλες ε, οδηγίες. Υπάρχουν ε, θέματα ε, τα οποία δημιουργούν προβλήματα, υπάρχει επισφάλεια για τους πολίτες, είναι πολύ σκοτεινές οι διάφορες πρακτικές και υποθέσεις των τραπεζών. Η τράπεζες προσπαθούν να μην εφαρμόσουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αρνούνται όλες τις επιτυχίες μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τα οποία μπορεί να προστατεύσουν τους πολίτες ε, για αυτές τις πρακτικές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις και ο τραπεζικός τομέα έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα κοινωνικής επισφάλειας ε, για να εκμεταλλευτούν πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες βρίσκονται πλέον σε δύσκολη κατάσταση. Δεν ε, λύνονται τα προβλήματα, οι ε, μισθοί είναι αναξιοπρεπείς, υπάρχει ενεργειακή ένδια και ένδια των παιδιών. Απόλυτη δηλαδή φτώχεια στον 21ο αιώνα και μάλιστα στην Ευρώπη των ευκαιριών. Εμείς ε, δίνουμε μάχη λοιπόν ε, κατά αυτών των θεμάτων στους δρόμους μαζί με τις οικογένειες. Ε, εξετάζουμε και την ομοθεσία και των οικονομικών αγορών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βοηθούμε τις οικογένειες για να περάσουν στις διαδικασίες για τις υποθήκες για να ανακτήσουν τις κατοικίες τις οποίες έχασαν. Προσπαθούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τις οικογένειες να αποκτήσουν μια νέα ζωή μετά από τις πολιτικές που εφαρμόζονται που τις έχουν ξεχάσει ε, αυτοί που έκαναν την οικονομική προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα ασφάλματα τα οποία έχουν διαπράξει οι τράπεζες και είναι αυτές οι οποίες χρειάζονται να κάνουν τη μεγαλύτερη προσπάθεια. Εδώ και ένα χρόνια ξεκίνησε μια διαδικασία ε, προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και ε, γι' αυτό ακριβώς επειδή δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τις ε, αποφάσεις ε, ζητήσαμε ε, μέσω της αναφοράς αυτής ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εφαρμόζει καλύτερη διαφάνεια στα προγράμματα υποθηκών ε, και για το δημόσιο και για το ιδιωτικό χρέος. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές δυσκολίες να λάβουμε πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το πώς γίνονται αυτές οι συναλλαγές και πού προορίζονται αυτές οι επενδύσεις και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από ιδιωτικές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Ε, τα πάντα γίνονται με πολύ και καλυμμένο τρόπο ε, και αυτό είναι εις βάρος των οικογενειών οι οποίες πλήττονται από αυτή τη διαδικασία. Ζητούμε λοιπόν μια διαδικασία διαβάνειας να μας δείσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όλες τις πληροφορίες για τις επενδύσεις και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που έχουν κάνει και που έχουν πουλήσει αυτές τις επενδύσεις. Και επίσης δεν ξέρουμε καν σε ποιον έχουν πουληθεί όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε ε, τον κόσμο από τις ε, ε, ατασταλίες της Ισπανικής Τράπεζας. Ε, ε, πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι μπορούν να είναι όλοι πιστωτές. Θέλουμε να αποφύγουμε μια άλλη υπόθεση ε, υποθηκών έκπληξη. Εμείς οι πολίτες λοιπόν είμαστε αυτοί οι οποίοι πληρώνουμε όλα τα θεσμικά όργανα με τους φόρους μας, ακόμα και αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να ξέρουμε πού πάνε αυτά τα χρήματα και πού πάνε οι προσπάθειες των πολιτών, ανδρών και γυναικών. Θέλουμε λοιπόν να προχωρήσει η προσπάθειά μας. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω εγώ προς την ίδια κατεύθυνση. Όπως είπε και η συνάδελφος, θέλουμε από την Επιτροπή σας να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τηρήσει τα του κανονισμού της και να καταφέρουν όλοι οι πολίτες, όχι μόνο οι Ισπανοί, αυτοί οι οποίοι πλήττονται από αυτές τις τραπεζικές συναλλαγές, να έχουν, μπορούν ε, να προσφύγουν στο δικαστήριο κατά των τραπεζών. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα στη διάρκεια της κρίσης που βιώνουμε και σήμερα ξέρουμε τι γίνεται με αυτέ τις ε, υποθήκες. Υπάρχουν ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους. Παλιά υπήρχαν αποθεματικά και τώρα εμπιστοσύνη στι αγορέ. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οι οικονομικές αγορές όμως πλέον ε, κάνουν κερδοσκοπικές συναλλαγές και ε, επομένως και οι εθνικές ε, τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και τα ευρωπαϊκά θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες πάγιες πρακτικές και να εφαρμόζεται νομοθεσία που έχει εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να είναι δημόσια και προσβάσιμα όλα αυτά και να τηρούνται οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί επί των θεμάτων. Με τα προγράμματα αγοράς δημοσίου και ιδιωτικού εισαγοράς ε, χρέους έχουν ε, δημιουργήσει ε, ύποπτε συναλλαγέ και αγοράζουν οι ίδιοι όλα τα προβληματικά προϊόντα και μας έχουν οδηγήσει σε μια καταβόθρα χρέου. Επομένως πρέπει να, βρούμε, να δούμε τι θα κάνουμε για να μπορέσουμε να προσφύγουμε κατά των τραπεζικών αρχών και να μπορέσουμε να προστατεύσουμε χιλιάδες πολίτε. Πρέπει να υπάρχουν πιο μόνιμες λύσεις, διότι προσπαθούν να παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν λιγότεροι στις υποθέσεις τους. Υπάρχει και το Συνδικάτο των ε, Μετόχων, που είναι το Συνδικάτο αυτό το οποίο ε, υπερασπίζεται αυτούς τους ανθρώπους που ε, παίρνουν χρήματα από τις υποθήκες. Διαγράφεται όμως η προστασία προς τους επενδυτές και δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορέσει να ζητήσει απολογισμό για τα όσα συμβαίνουν. Υπάρχουν λοιπόν ε, επιχειρήσεις διαχειριστών Σε su Real Decreto 2015 από το 2015 λοιπόν δίνονται αυτά σε ε, εταιρείε διαχειριστών και πρέπει να ξέρετε ότι αυτές οι επιχειρήσεις ε, στην πλειοψηφία τους είναι ιδιοκτησία των τραπεζών. Επομένως είναι όλα και καλυμμένες υποθέσεις. Πλήττονται λοιπόν όλοι όσοι έχουν ένα υπόθηκο δάνειο αλλά ακόμα και θεσμικοί επενδυτές. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι χάνουμε τα ωφέλη και δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ε, πίσω από κάθε ενεργητικό, όπως ε, αποκαλούν τις υποθέσεις μας, ε, υπάρχει μια οικογένεια που έχει βρεθεί στο δρόμο λόγω αυτής της αδικίας. Όταν μπορέσουμε να επαληθεύσουμε πώς οι Ισπανικές τράπεζες έκαναν όλη αυτή την υπόθεση, καταφέραμε ότι πρέπει να προσφύγουμε για να μπορέσουν να σταματήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες υποθηκών γιατί ε, το πρόβλημα είναι ότι οι τράπεζες δεν είναι ιδιοκτητές αυτών των ενυπόθηκων δανείων στην πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τα στοιχεία λοιπόν και τα ζητούμε εμεί μέσω τη αναφορά μα. Υπάρχει υποχρέωση να γίνεται τακτική ενημέρωση για την εξέλιξη των κονδυλίων και τι γίνεται με τι διανοδοτήσει και γι' αυτό ακριβώ και ζητούμε και εμεί ε, να δίνονται αυτά τα στοιχεία. Ε, θα μπορούσαν μέσω μια αναφορά να μα πούνε σε ποιο ταμείο βρίσκεται τον υπόθηκο δάνειών μα. Εμεί ζητούμε το δικαίωμα στην ε, ενημέρωση για να υπερασπιστούμε τα σπίτια μα και τι οικογένειέ μα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλέσω ε, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο, τον κύριο Έρχαρτ και τον κύριο Σπηλέδας Μάρτος. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριο Σέρχαρτ. Ακούσαμε πολλές πτυχές. Εγώ θα περιοριστώ ε, στο θέμα της αναφοράς. που είναι το, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η υποχρέωση ε, του Ισπανικού Οργανισμού Τυπλοποίησης να οργανώσει ένα αποθετήριο των πληροφοριών και να δίνει πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα που έχουν αγοράσει. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να δημοσιεύονται. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι αναφέροντες ζητούν τις πληροφορίες αυτές ώστε μετά από την παροχή δανείου να ε, μπορούν να γνωρίζουν τα περί του δανείου και να μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ε, στα δικαστήρια. Και ε, υπάρχει ένα θέμα στην αναφορά το οποίο δεν έχω καταλάβει απόλυτα. Ε, οι αναφέροντες ε, πάντως πολύ σωστά είπαν ότι ήδη έχουν αναφέρει το θέμα αυτό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Και οι δύο απάντησαν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει τη δυνατότητα να παρέχει τις πληροφορίες αυτές Δυστυχώ για του αναφέροντες ε, και εγώ καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα και θα σας εξηγήσω σύντομα γιατί. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι δημόσιος οργανισμός. και έχει εποπτικά καθήκοντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στον κανονισμό που έχει να κάνει με τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ε, προχωρήσει πέρα από τις αρμοδιότητες αυτές. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αρμόδια ε, για την προληπτική εποπτεία των τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Δεν είναι λοιπόν αρμόδια για τα ε, ισπανικά ε, ταμεία υποθηκών ε, ή για την τιτλοποίηση. ο ισπανικός οργανισμός εποπτείας είναι αρμόδιος για τα ταμεία αυτά και σύμφωνα με τον κανονισμό για τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι ε, ο υπερεπόπτης. Από ό,τι κατάλαβα, οι αναφέροντες θέλουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ζητήσει από τον ε, Ισπανικό Εποπτικό Οργανισμό να κάνει κάτι. Αυτό όμως μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μόνο για τις τράπεζες, όχι όσον αφορά την τιτλοποίηση. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Αυτό δεν ε, εμπίπτει στι αρμοδιότητε ε, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπω κάθε δημόσιο ε, φορέα, πρέπει να παραμένει εντό των αρμοδιοτήτων που τη παρέχει ο νόμο. Τούτου λεχθέντος και έχοντας ακούσει αυτά που μόλις είπαν οι αναφέροντες, Ανέφερε ότι θέλουν να γνωρίζουν πού καταλήγει το ενυπόθηκο δάνειο, εάν πολιθεί σε ποιον πωλείται και υπό ποιες προϋποθέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που ρυθμίζεται κυρίως στο αστικό δίκαιο, είναι δηλαδή θέμα των εθνικών νομοθετών. Εκτός από πολύ περιορισμένο αριθμό υποθέσεων, ο ευρωπαϊκός νόμος λοιπόν εδώ πέρα δεν μπορεί να αποτελέσει προσανατολισμό. Όσον αφορά το δεύτερο αίτημα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αποκαλύψει πληροφορίες ε, πάνω στα προϊόντα που έχει αγοράσει στον τομέα αυτών, προς όφελος όσων επηρεάζονται των ε, ε, ιδιωτών καταναλωτών δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πάλι πρέπει να ενεργεί στο πλαίσιο των κανόνων που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν όταν αγοράζει αυτά τα προϊόντα τα αγοράζει επίσης όρις με οποιονδήποτε τρίτο. Δεν έχει λοιπόν ε, αυξημένη υποχρέωση να δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση στο θέμα αυτό και η δεύτερη είναι ότι μάλλον ε, θα παραβιάζει και τις ε, διατάξεις ε, για την προστασία των δεδομένων εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύσει τις σχετικές πληροφορίες, διότι Ε, όλες οι πλευρές ε, στη συναλλαγή αυτή έχει δικαίωμα για προστασία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν δεν έχει ε, τη δυνατότητα, δεν έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές. Συνοψίζοντας λοιπόν, δεν υπάρχει νομική βάση για αποκάλυψη από πλευρά πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας των πληροφοριών αυτών, ούτε υπάρχει νομική βάση ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να καλέσει την ε, Ισπανική Εποπτική Αρχή να δημοσιεύσει τις πληροφορίες. Και μια τέτοια νομική βάση θα ήταν απολύτως απαραίτητη για να μπορέσει να ενεργήσει νόμιμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να κάνει αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δίνω το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω καταρχάς τους ε, ε, φίλους από την Ισπανία που έχουν θέσει όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι δύο θέματα, θα έλεγα, διαφορετικά. Το ένα έχει να κάνει με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως επενδυτή και ως εποπτική αρχή. Και το δεύτερο είναι τα ε, NPLs όπως λέμε, τα κόκκινα δάνεια, το οποίο είναι ενδιαφέροντος για όλους μας. Καταρχάς έχουμε πει αρκετές φορές και εγώ προσωπικά ότι υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία είναι υποτίθεται ανεξάρτητη νομισματική αρχή είναι εποπτική αρχή των συστημικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρα το 80% των τραπεζών το ελέγχει, τις μεγάλες τράπεζες ελέγχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επομένως και τις μεγάλες ισπανικές τράπεζες, είναι μέλος της Τρόικας και ασκεί πολιτική στα κράτη-μέλη που ήταν με μνημόνιο και είναι και επενδυτής διότι αγοράζει επενδυτικά προϊόντα. Δεν μπορεί ο κύριος Ντράγκη να φοράει τέσσερα καπέλα ταυτόχρονα. Δεν γίνεται. Είναι σε σύγκρουση συμφερόντων. Και αυτό το έχουμε πει και στην Επιτροπή μας εδώ, αλλά και στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Όταν λειτουργεί στο, στην ποσοτική χαλάρωση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες τι κάνουν. Αγοράζουν δημόσιο χρέος και αγοράζουν ιδιωτικό χρέος. Έχω ρωτήσει επανειλημμένα τον κύριο Ντράγκη να μας πει πληροφορίες για το πώς αγοράζει δημόσιο και ιδιωτικό χρέος η Τράπεζα τη Ελλάδο. Η τράπεζα της, ε- ενώ η Ελλάδα Φερρυπίν δεν είναι στην ποσοτική χαλάρωση, η τράπεζα της Ελλάδος μέχρι σήμερα το 2015 και 2016 έχει δώσει 42,5 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει συμμετάσχει στην ποσοτική χαλάρωση. Το πρώτο που ρώτησα είναι που βρήκε τα λεφτά. Το δεύτερο είναι τι ομόλογα έχει αγοράσει. Και δεν απαντούσε. Έδινε γενικές απαντήσεις. Τον ρώτησα σε ποιες ιδιωτικές επενδύσεις έχει μπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τι ομόλογα έχει αγοράσει. Αν έχει αγοράσει η Deutsche Bank, η οποία ήταν σε πρόβλημα επί ένα διάστημα. Είπε ο κύριος Δράγκη, δεν σας δίνω αυτές τις πληροφορίες, γιατί λέει θέλει να προστατεύσει τους επενδυτές. Αλλά εγώ ρωτάω, πώς θα ξέρουμε εμείς ποιες εταιρείε πραγματικά βοηθούνται μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης διότι υπήρχαν καταγγελίε ότι στην Ισπανία η, Ευρωπα... η Κεντρική Τράπεζα τη Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν αγοράσει ομόλογα μόνο πέντε μεγάλων ισπανικών εταιριών και από καμία άλλη. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρξει διαφάνεια. Δεν πρέπει να δούμε το θέμα αυτό. Στην Ελλάδα η Τράπεζα της Ελλάδος με απάντηση γενικόλογη του κυρίου Ντράγκη αποδείχθηκε ότι έχει αγοράσει ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων η οποία μετά δανειοδότησε τη Φραπόρτ, η οποία μετά Φραπόρτ άρπαξε τα 14 ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια. Έδωσε, αγόρασε ομόλογα η Τράπεζα της Ελλάδος, η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, από το θέμα του ESM, και μετά ο ESM επέβαλε μνημόνιο στην Ελλάδα δίνοντα δανεικά. Αυτά είναι εξωφρενικά που συμβαίνουν. Και δεν συμφωνώ με αυτά που μα λέει η Κομισιόν. Όλα πρέπει να έρθουν στο φω. Να δούμε πώ διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπω και η Κεντρική Τράπεζα τη Ισπανία, όπω και η Κεντρική Τράπεζα τη Ελλάδο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ιδιωτικό χρέο, τα NPLs. Διότι πολλούνται αυτά τα δάνεια και πολλούνται αντί πινακίου φακής και τα αγοράζουν αυτά τα δάνεια τα κοράκια και εν συνεχεία πηγαίνουν και κάνουν έξωση, αρπάζουν τα σπίτια. Έχουμε δει απίθανε εικόνε και σκηνέ στην Ισπανία να πετάνε ηλικιωμένους έξω από τα σπίτια και φοβάμαι ότι θα δούμε αντίστοιχα θέματα και στην Ελλάδα τώρα που επιτρέπονται οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Επομένω, δεν μπορεί να πουλά απλά ένα δάνειο, να το τίτλοποιεί και ο δικαιούχο, ο, δανει, ο, να μην γνωρίζει ποια είναι η τύχη του δανείου του για να μπορεί να, έχει, να παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη και συμβαίνουν επίσης απίθανα πράγματα διότι οι τράπεζες οι ιδιωτικές στην Ισπανία πήραν 50 δισεκατομμύρια ευρώ για να διασωθούν. Στην Ελλάδα πήραν πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιο έδωσε αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα στην ουσία έχουν χρεωθεί στον Ισπανικό λαό και στον ελληνικό λαό. Και έχουν υποστεί μνημόνια και μέτρα περιοριστικής πολιτικής και μείωση συντάξεων και μισθών. Επομένως, δεν είναι αυτό που λέγεται από την Κομισιόν ότι δεν θα δίνει καμιά ενημέρωση, καμία τράπεζα του πού πήγαν τα χρήματα και πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα κόκκινα δάνεια, αν έχουν πουληθεί στα funds, τα επιθετικά, τα distress funds, τα κοράκια. Και μάλιστα αντίπεινα και ουφακής. Τέλος, υπάρχουν απαντήσεις και λύσεις. Διότι στην Κύπρο υπάρχει μια ρύθμιση σωστή που λέει Εάν μια τράπεζα πουλήσει το δάνειο ενός ιδιώτη, έστω ότι το δάνειο είναι 100.000 ευρώ στεγαστικό δάνειο και το πουλήσει σε distress fund η τράπεζα σε 3.000 ευρώ, οφείλει να καλέσει το δανειολήπτη να πει αν μπορεί να δώσει 3.000 ευρώ να αγοράσει αυτό το δάνειό του. Και αυτή είναι η σωστή πρακτική, την οποία δεν εφαρμόζουν στην Ελλάδα και είδα ότι δεν εφαρμόζουν και στην Ισπανία. Υπάρχουν λοιπόν λύσεις, υπάρχουν απαντήσεις. Εμείς έχουμε προτείνει τη δημιουργία ενός Ταμείου Διάσωσης των Δανειοληπτών στην Ελλάδα, ένα ταμείο το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί με 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το υπόλοιπο δάνειο που πήρε η Ελλάδα με το τρίτο δανειακό πακέτο και να μπορεί ο δανειολήπτης να πάει να αγοράσει το δάνειό του στην τιμή πρώτης προσφοράς που θα δοθεί το, στο Distress Fund. Υπάρχουν λοιπόν προτάσεις, αλλά το θέμα είναι πολιτικό κυρία Πρόεδρε. Δεν επιθυμεί σήμερα η τραπεζοκρατία να δώσει λύσεις. Και τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ταγιάννη, ο οποίος προχτές έστειλε κυρία Πρόεδρε μία επιστολή στον κύριο Ντράγκη και διαμαρτύρεται για την πολιτική της ΕΚΟΥΤΟΥ διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχτές αποφάσισε νέους κανόνες υπό τους οποίους οι τράπεζες θα εξεφορτωθούν τα κόκκινα δάνεια. Τελειώνω. Και υποχρεώνει τις τράπεζες να εγγράψουν μέσα στους ισολογισμούς τους εντός μιας εφταετίας τα δάνεια που είναι καλυμμένα με υποθήκες και εντός μιας διετίας τα δάνεια που είναι καταναλωτικά. Και ορθώς είπε ο κύριος Σταγιάννη ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφασίσει μονομερός ο κύριος Δράγκη. Και ορθώ είπε ο κύριο Σταγιάννη και νομίζω ότι εκφράζει όλου μα και όλου σα και εσά, κυρία Πρόεδρε, ότι το θέμα αφορά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι συνομοθέτης και στην επιστολή του ο κύριος Ταγιάννη λέει στον κύριο Ντράγκη ότι αν συνεχίσει αυτή την τακτική η κεντρική τράπεζα θα οδηγήσει σε διαθεσμική κρίση, interinstitutional crisis, διότι έχει αρμοδιότητα το κοινοβούλιο μας να δει τις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια. Επομένως, κλείνοντας, θεωρώ απαράδεκτο το ότι δεν έχει έρθει εδώ η κεντρική τράπεζα. Οφείλει να έρθει εδώ να τοποθετηθεί. Και από εκεί και πέρα εμείς εδώ προτείνω πρώτον να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά οπωσδήποτε, να ενημερώσουμε την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, να ενημερώσουμε προσωπικά τον κύριο Ταγιάννη, γιατί νομίζω ότι αυτή η αναφορά συμβαδίζει με την επιστολή που έστειλε προς τον κύριο Ντράγκη και να ζητήσουμε να έρθει εδώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι οφείλει να δώσει απαντήσεις είναι ο πιο ισχυρός οργανισμός, είναι, ανεξέλεγκτη αρχή, είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά δεν είναι ανεξέλεγκτη αρχή. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει. Ευχαριστώ. κυρία Ευχαριστώ. Είναι αλήθεια ότι το πρόβλημα της στέγασης ε, στην Ισπανία είναι πάρα πολύ σοβαρό και προγαλεί πραγματικές ε, τραγωδίες. Άνθρωποι μένουν χωρίς σπίτια, ε, οικογένειες που βλέπουν τις οικονομίες τους και τις προσπάθειες μιας ζωής να εξανεμίζονται και ε, είχαμε και ανθρώπους που αυτοκτόνησαν λόγω της, του δράματος αυτού των χρεών. Ε, η βασική ευθύνη είναι για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά τουλάχιστον ελπίζαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστήριζε τους ε, ε, Ευρωπαίους πολίτες και όχι αυτές τις αγορές, τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Και η αλήθεια είναι ότι μας εξέπληξε ιδιαίτερα η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι καταρχάς μας είπε ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μετά στη συνέχεια μα είπε ότι ούτε τη Κεντρική τράπεζα είναι η ευθύνη. Ουσιαστικά ήταν ένας κομψός τρόπος να μας πει ότι η αρμοδιότητα γι' αυτό δεν είναι κανενός. Κάτι το οποίο με παρεξενεύει, διότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία για το δικαίωμα ενημέρωσης του καταναλωτή είτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιος από τους δύο έχει ευθύνη να τηρηθεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενημέρωση στους καταναλωτές. Και αν κάποια χώρα δεν τηρεί τις προϋποθέσεις διαφάνειας και της ενημέρωσης προς τους ε, καταναλωτές, να υπάρξουν μια διαδικασία επιπαραβάση και να, να επιβληθούν κυρώσεις. Και κάποιο πρέπει να το κάνει αυτό. Τώρα, ποιανού είναι η ευθύνη δεν ξέρω, ή τη Κεντρική Τράπεζα ή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι φταίει περισσότερο η Επιτροπή. Υπάρχει υποχρέωση διαφάνεια ενημέρωση και αυτό ζητούν και αναφέροντε. Οι αναφέροντε, αν κατάλαβα καλά, δεν ζητούν καν να μην πουληθούν ε, οι υποθήκες τους ε, σε άλλα ταμεία. Ζητούν απλώς να τους δώσουν πληροφορίες για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ε, του ενυπόθηκου δανείου τους, γιατί έτσι γνωρίζοντας ποιος είναι ο ιδιοκτήτης μπορούν να αποφύγουν τη χρεοκοπία και τους πληστηριασμού. Μπορεί να αποφύγουν να μείνουν άνθρωποι στους δρόμους, σε ολόκληρε οικογένειε. Και νομίζω λοιπόν ότι σίγουρα υπάρχει ευθύνη, σίγουρα υπάρχει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει να τηρηθεί ε, η οδηγία και επομένω εδώ απευθύνομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι οδηγίε για να τηρούνται αλλιώ πρέπει να έρθει σε επαφή με την Ισπανική κυβέρνηση. Και το άλλο το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω και την ε, πρόεδρο της Επιτροπής είναι κατά πόσον έχουμε τη δυνατότητα εμείς ως ε, ε, Επιτροπή Αναφορών να αποτανθούμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό, να απευθυνθούμε σε αυτούς για να εκθέσουμε την κατάσταση, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση προς τους χρήστες για το ποιος είναι ο, ο κάτοχος των τίτλων της υποθήκη τους και να μπορέσουμε να διαβιβάσουμε αυτές τις ανησυχίες προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νομίζω ότι και αυτός είναι ένας τρόπος να δράσουμε. Αντί να απευθυνθούμε απλώς στις Ισπανικές Αρχές και να μας πούνε γιατί δεν τηρούν τις ευρωπαϊκές οδικίες ε, για την υποχρέωση ενημέρωση προς καταναλωτές. Επίσης, ε, αν συμφωνεί και ο συνάδελφο, αν ε, συμφωνεί και η πρόεδρο και αν συμφωνούν και αναφέροντες, ίσω ε, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αυτέ τι δύο οδού. Δηλαδή, να αποτανθούμε προ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και να έρθουμε και σε επαφή με τι Ισπανικέ αρχέ για να μάθουμε ε, ή μάλλον να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία και θα ήθελα να ξέρουμε γιατί δεν υπάρχουν πληροφορίες για τους καταναλωτές. Ε, για μένα αυτή είναι η κατάλληλη πρόταση. Αυτά ευχαριστώ. Εξαιρετικά. Οι αναφέροντες θέλουν να προσθέσουν κάτι μετά από όσα άκουσαν από τους συναδέλφους. Παρακαλώ. Ναι. Νομίζω ακούσαμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαφωνούμε με όλα όσα ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τίποτα δεν συμφωνούμε. Ε, δεν ξέρω, ή δεν τα είπαμε εμεί σωστά, ή δεν τα μα καταλάβανε καλά, δεν καταλάβατε το χαρακτήρα τη αναφορά. Η αναφορά βασίζεται σε μια ευρωπαϊκή οδηγία, την 24 του 2013. Εκεί έχουμε τα πάντα όσον αφορά την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και σε αυτό τον κανονισμό, τον 1024 του 2013, πέραν ε, το θέμα της εποπτείας ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υπάρχει και μια σειρά από διατάξεις που καλύπτουν το θέμα μας. Και σε αυτό τον, ε, την οδηγία υπάρχει και το θέμα της συνεργασίας με την ε, Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας για την ε, προστασία των καταναλωτών. Επίσης, αυτό το οποίο σας λέμε εμείς σήμερα ήδη έχει γίνει πριν από μερικά χρόνια από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν ε, κατάρτισε τον κανονισμό και ζήτησε από την Τράπεζα της Ισπανίας να δημοσιεύσει τα στοιχεία των ε, ε, υπηρεσιών τιτλοποίησης, των επιχειρήσεων τιτλοποίησης και να έχει ένα παράρτημα με όλες τις τιτλοποίησεις και τα στοιχεία ενεργητικού που τιτλοποιήθηκαν και όμως ε, η Επιτροπή Διαχείρισης ε, και ε, το Οργανισμός Τιτλοποίησης έχουν στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πρόκειται για φωτοτυπίες, για χιλιάδες υποθήκες τις οποίες δεν μπορούμε να μελετήσουμε έτσι όπως μας τις δίνουν. Το μόνο λοιπόν που ζητάμε είναι να τηρήσετε τα όσα προβλέπει ο κανονισμός, να τηρήσετε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που διέπει αυτό. 1024 του 2013 σε όλες τις διατάξεις και την προστασία των καταναλωτών που αναφέρεται στο άρθρο 29. Και πέραν των επιχειρημάτων που ήδη εκθέσαμε στην αναφορά μας, που περιλαμβάνει πολύ σημαντικά επιχειρήματα και όλα έχουν σχέση με το σχετικό κανονισμό, όπως για παράδειγμα το άρθρο 3 που αναφέρεται στη συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά όλων των αρμοδίων αρχών ε, της κεφαλαιογοράς, ε, της ε, αρχές επενδύσεων κλπ. κλπ. το 57 που αναφέρεται στο δικαίωμα του Κοινοβουλίου να συστήσει επιτροπή για να ρυθμίσει τα πάντα ε, επί του θέματος. Ε, δεν αναφερόμαστε λοιπόν σε πάυση πληρωμών ή σε δικαστήρια ή σε οτιδήποτε άλλον. Εμείς απλώς κυρίως λέμε ότι παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης, κυρίως το άρθρο 42 για το δικαίωμα σε πρόσβαση σε έγγραφα και επίσης ε, το 48 τη βοήθεια προς τους καταναλωτές και το δικαίωμα στην ενημέρωση που δεν ε, ε, περιλαμβάνονται στα στοιχεία που μας στέλνει η Επιτροπή και μας φαίνεται ακατανόητο ότι η πρώτη απάντηση της Επιτροπής λέει ότι ο Ευρωπαίος ρυθμιστής είναι ένας ακόμα αγοραστής ενώ είναι αυτός ο οποίος θα έπρεπε να φροντίζει τη βιωσιμότητα του συστήματος της, ε, των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητούμε λοιπόν να παραμείνει αναφορά όπως είπαν και οι ευρωβουλευτές προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το οποίο κάναμε με τη συγκεκριμένη αναφορά. Πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Ήρθαμε σε επαφή με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και ζητήσαμε τη γνωμοδότησή τους. Έχω την απάντηση και νομίζω ότι την έχετε κι εσείς. Έχει διανεμηθεί στην αίθουσα και θα ήθελα να σας τα διαβάσω. Ένα τμήμα της απάντησης της ΕΚΟΝ λέει ότι από τότε που συνετάχθη η αναφορά έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις σε σχέση με την τιτλοποίηση και την προστασία των συμφερόντων των αναφερόντων. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσαν ένα ανεπίσημο τριμερή διάλογο έτσι ώστε να υπάρξει ένας κανονισμός για την τυπλοποίηση το ταχύτερο δυνατόν που να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των αναφερόντων. Αυτή τη στιγμή στεθεί το έγγραφο αυτό σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2019. Ε, το κείμενο το οποίο έχει καθοριστεί είναι σε προσωρινή ακόμα βάση διατύπωσης, αλλά ελπίζουμε να περιλαμβάνει τις εξής καινοτομίες. Πρώτον, αυξημένη διαφάνεια και απαιτήσει διαφάνειας οι οποίες θα ξεπερνούν αυτά τα οποία προβλέπει το 34 του Ισπανικού νόμου 5 Η δημιουργία μιας αγοράς τιτλοποίησης όπου οι συμμετέχοντες στις αγορές και οι αρμόδιες αρχές θα είναι σωστά ενημερωμένες για όλες τις διαδικασίες τιτλοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και κατά μεμονωμένο δάνειο, κατά περίπτωση. Λοιπόν, το υπογράφει ο συνάδελφος Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη και με αυτό, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε κύριε Μαριά. Να μου επιτρέψετε να κλείσω ή θέλετε να, να μιλήσετε πριν κλείσω το θέμα. Θα κρατήσουμε λοιπόν ανοιχτή την αναφορά αυτή και θα επανέλθουμε με μια επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνοδευόμενη από την γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΚΟΝ και θα προσπαθήσουμε με ευγένεια να διευρύνουμε την πρόσκληση και σε μια συνάντηση και με τις άλλες επιτροπές. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν θα είναι όλοι παρόντες. Ελπίζω ότι είναι καλό να είναι κανείς ευγενής. Ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεσμεύεται από τον κανονισμό λειτουργίας της, αλλά εμείς θα πρέπει να τους δείξουμε ότι τις αναφορές θα πρέπει να τις λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά και όπως πρότεινε άλλωστε και η ίδια η κυρία Αλμπιόλ θα επανέλθουμε στο θέμα της επαφής με τις Ισπανικές Αρχές θα τους δώσουμε αντίγραφα των επιστολών και των γνωμοδοτήσεων. Κύριε Μαριά, τι προτιμάτε να κάνουμε. Καταρχάς συμφωνώ με την τοποθέτησή σας ότι πρέπει να αποσταλεί η επιστολή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμως, επειδή προκύπτει από την απάντηση του κυρίου Γκαλτιέρη ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία φάση διαβούλευσης Πιστεύω ότι θα πρέπει να έρθει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναγίνει συζήτηση επί του θέματος, να έχουμε και τους petitioners για να καταλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι και αυτή ελέγχεται. Ελέγχεται κατά την έννοια από τους πολίτες. Δεν είναι ένα όργανο ανεξέλεγκτο. Πιστεύω λοιπόν ότι ερχόμενοι εδώ σε μια δημόσια συζήτηση με live streaming να δεσμευτεί σε απόψεις όχι πίσω από κλειστές πόρτες και ενημερώσεις. Εδώ λοιπόν μπροστά στους πολίτες, οι πολίτες την καλούν μέσω βεβαίως του Κοινοβουλίου μας, αλλά εδώ θα είναι και οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές και οι ετούντες, γιατί όπως βλέπετε παρακάτω υπάρχουν και άλλοι που διαφωνούν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, να μπουν τα θέματα στο τραπέζι και να δεσμευτούν ότι θα πάρουν τέτοιες αποφάσεις που θα είναι υπέρ των πολιτών και όχι υπέρ των κολλητών, δηλαδή υπέρ των τραπεζών. Αυτό να είναι σαφέστατο. Από εκεί και πέρα συμφωνώ με τις προτάσεις σας. So, we do that. And with that I... Αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μέχρι τις Βρυξέλλες. Ε, καλή επιστροφή σας εύχομαι. Και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στο θέμα αυτό, στο μέτρο που είναι δυνατόν. Να προχωρήσουμε τώρα στην επόμενη αναφορά, υπαριθμόν 91 του 2013 που επίση έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη διαφάνεια. Δεν είναι παρόν ο αναφέρον, είναι παρούσα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δίνω λοιπόν ε, τον λόγο ε, στον κύριο Σεβαστιάν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την Επιτροπή σας που δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει τις θέσεις της ε, για το θέμα αυτό. Ε, έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δώσει πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό και το προσωπικό της και τις οικονομικές συναλλαγές μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια. Επίσης, ζητάει ο αναφέρον από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δημοσιεύσει τα ονόματα των δικαιούχων και τα ποσά των συναλλαγών αυτών. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε το 2012 και τον Μάρτιο του 2014 και απάντησε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να ε, διεξάγει συναλλαγέ ε, για λόγου του προσωπικού της. Αυτό δηλαδή είναι σύμφωνο με ε, τη συνθήκη. Ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απήντησε ότι δεν είναι σε θέση να δημοσιεύσει τις πληροφορίε που ζητάει ο αναφέρον. Καλούμε τον αναφέροντα ε, να απευθυνθεί ε, απευθεία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι εσωτερικό θέμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι παρατηρήσεις που είχαμε υποβάλει τότε ισχύουν και σήμερα και θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο του 2012 ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητής ε, σημείωσε ότι σωστά η Ευρωπαϊκή ότι ήταν σωστή απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στον αναφέροντα, ο αναφέρον καλείται να ζητήσει πιο συγκεκριμένε πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εφόσον δεν είναι παρόν ο αναφέρον, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο. Έχει ανακύψει, με αφορμή αυτή την ε, αναφορά, είναι τι κατάσταση επικρατεί στον τομέα των προσλήψεων από πλευράς ΕΚΤ. Διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα όργανα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προχωρεί σε μόνιμες προσλήψεις με το σύστημα των φωνξιονέρ που γνωρίζουμε, με δημόσιους διαγωνισμούς και κατά κύριο λόγο, σύμφωνα και με πολλά δημοσίευματα, διότι δεν έχουμε πληροφορίες, αρκείται στο να κάνει προσλήψεις προσωρινές, δύο-τριών ετών συμβάσεις, τεσσάρων ετών και δεν υπάρχει καθόλου διαφάνεια. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε επιπλέον πληροφορίες διότι θέλουμε να ξέρουμε υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποια κριτήρια προσλαμβάνονται τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα οποία αυτή τη στιγμή παίρνουν κολοσιαίες αποφάσεις για την Ευρώπη. Διότι ας το ξεκαθαρίσουμε αυτή τη στιγμή το ισχυρότερο, δυστυχώς, το ισχυρότερο θεσμικό όργανο σε όλη την Ευρώπη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι αποφάσεις που παίρνει επηρεάζουν τις τράπεζες, επηρεάζουν τους πολίτες, επηρεάζουν την ανεργία, επηρεάζουν τη φτώχεια. Δεν μπορεί λοιπόν χωρίς όρους και προϋποθέσεις να έχει ένα σύστημα προσλήψεων ιδιαίτερα κλειστό, χωρίς να υπάρχει διαφάνεια, χωρίς να γνωρίζουμε και από εκεί και πέρα πάμε στο δεύτερο θέμα. Τι γίνεται με το σύστημα των revolving doors Δηλαδή όσοι είναι στελέχη της ΕΚΟΥΤΟΥ υπό ποιου όρους και προϋποθέσεις δεσμεύονται ούτω ώστε μετά να μην πάνε να εργαστούν σε ιδιωτικές τράπεζες τις οποίες υποτίθεται ελέγχουν. Άρα λοιπόν το θέμα παρότι ο αναφέρον δεν είναι εδώ ίσως δεν είχε και τη δυνατότητα την οικονομική να έρθει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά, να συζητήσουμε και με μια κάποια άλλη επιτροπή του, ε, του Κοινοβουλίου μας για να δει το θέμα αυτό, διότι πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Έχουν γίνει πολλές καταγγελίες σε εφημερίδες και νομίζω ότι το θέμα της οργάνωσης και των υπηρεσιών της ΕΚΤ και του τρόπου προσλήψεων και των αμοιβών και των παροχών και των ε, ε, incompatibilities που πρέπει να έχουν, νομίζω ότι όλα πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Ευχαριστώ. more operations mm. on transactions. Okay. Mm. So. Καλώς λοιπόν θα κάνουμε το εξής, θα κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή και θα ζητήσουμε για μια ακόμη φορά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ξεκαθαρίσει την απάντησή της. Η τράπεζα έχει κάνει ε, ε, στο όνομα των μελών της τραπεζικές δραστηριότητες, έχει κάνει τραπεζικές συναλλαγές προς όφελος του προσωπικού της και τίθεται το θέμα εδώ για την πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα και τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε να ψηφίσουμε σε λίγο καιρό στην Ολομέλεια. Αυτή τη στιγμή πάρουμε την απόφαση, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά προς το παρόν θα κάνουμε αυτό το οποίο είπα. Συμφωνείτε. Καλώς. Περνάμε στο επόμενο θέμα το οποίο είναι η πολιτική χαμηλών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 683 ο αναφέρον δεν είναι παρόν και του ζητώ να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις ένα θέμα αρκετά περίπλοκο και αυτό σας ευχαριστώ Πρόεδρε Ο αναφέρον διαμαρτύρεται για τα χαμηλά επιτόκια. Λέει ότι χρησιμοποιεί λάθος το μέσο καθορισμού των επιτοκίων, του ύψους των επιτοκίων, εις βάρος των καταθετών. Δημιουργούνται απώλειες στα περιουσιακά στοιχεία των καταθετών. Λέγει ότι θα πρέπει να αλλάξει η ρύθμιση αυτή για να ενισχυθεί η οικονομία η Επιτροπή ΕΚΟΝ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απάντησε στην Επιτροπή Αναφορών τον Απρίλιο του 2017 και εμείς θα συμφωνήσουμε με την γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Συμφωνούμε με την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Το θέμα αυτό, η αναφορά αυτή συνδέεται με τα προβλήματα της νομισματικής πολιτικής. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μία από τις αρμοδιότητες έστω και επιμέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό περιγράφεται στη συνθήκη στο άρθρο 130 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται στη συγκεκριμένη περίπτωση την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι υπόλογη όμως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για το ύψος των επιτοκίων και στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και στα πλαίσια του τακτικού νομισματικού διαλόγου με τον κύριο Ντράγκη και στα πλαίσια των εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας της Επιτροπής ΕΚΟΝ, όπως επίσης και μέσω προφορικών ερωτήσεων τις οποίες έχουν καταθέσει προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με μονομένα μέλη. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο άπτεται των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σαν ε, Επιτροπή ζητάμε από την δική σας Επιτροπή να στραφεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, η ε, τράπεζα απάντησε χθες, 10 Οκτωβρίου έχετε την απάντηση. Είναι μια μεγάλη επιστολή, λέει η Πρόεδρος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τονίζει ορισμένα στοιχεία τα οποία μπορούμε να δούμε τώρα πλέον. Η απάντηση στις γραπτές ερωτήσεις των βουλευτών από πλευράς των αντιπροέδρων οι οποίοι έρχονται ε, κάθε χρόνο στο Κοινοβούλιο για να παρουσιάσουν την ετήσια έκθεση ελήφθησαν μέτρα τον Ιούνιο του 2014 τα οποία οδήγησαν στην ποσοτική χαλάρωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται ασχολούνται με το θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει αλλά θα ήθελα να πω ότι αφού έχουμε διαβάσει την απάντηση αυτή αν και λίγο συνοπτικά θα... Κοιτάξτε κύριε Μαριά θα σας δώσω το λόγο πριν κλείσω τη συζήτηση γιατί μπορεί να καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Αν συζητούμε ταυτόχρονα και την, αναφορά 676 που είναι παρακάτω γιατί η απάντηση της Κεντρικής Τράπεζας έχει και τις δύο αναφορές. Ε, εάν συζητηθεί μετά, τότε θα μιλήσω μετά. I τότε θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφερθεί και στις ε, επόμενες δύο αναφορές για να τις ε, εξετάσουμε όλες μαζί. Και μετά θα αντιδράσει ο κύριος Μαριάς. Άλλοι συνάδελφοι δεν βρίσκονται στην αίθουσα. Λοιπόν, για να διευκολυνθεί η δουλειά θα ήθελα από την Επιτροπή να μας παρουσιάσει και τις δύο επόμενες αναφορές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η 0676 είναι αντίστοιχη με την προηγούμενη, διότι ο αναφέρον διαμαρτύρεται για πτυχές της νομισματικής πολιτικής και κυρίως ε, τα, επιτόκια τα οποία οδηγούν μικρές ε, σε μικρές επιστροφές για τους καταθέτες, κάτι το οποίο αναφέρθηκε ήδη, και μία ακόμα απόφαση που είναι η απόσυρση των ε, χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ. Ο αναφέρον ζητά να εγκριθεί νομοθεσία η οποία δεν θα επιτρέπει ε, την ε, καταστροφική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή θα βρει έναν τρόπο να απαντήσει σε αυτήν και ο ε, αναφέρον διαμαρτύρεται ότι η Γερμανία υποχρεώθηκε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρόπον την Α και στην Νομισματική Ένωση και να υπογράψει διάφορες συνθήκες. Ε, επί της ουσίας αναφέρθηκε ήδη ε, η η υπόθεση αυτή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η έκδοση χαρτονομισμάτων είναι συγκεκριμένη πολιτική ε, που είναι και πάλι αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για την νομοθεσία που ε, θα έπρεπε να απαγορεύει ή να απαντά στη νομισματική πολιτική ε, τότε αυτό δεν είναι εγγεγραμμένο στη συνθήκη και για το γεγονό ότι η Γερμανία υποχρεώθηκε να υπογράψει τη συνθήκη. εμει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε θεματοχύλακες των συνθήκων αλλά δεν παρεμβάνουμε για το κατά πόσον κάποιος θα υπογράψει ε, ε, ή θα υποχρεωθεί και αυτό νομίζω ότι δεν είναι και του πεδίου εφαρμογή. Ευχαριστώ. Ναι, νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλη συζήτηση από αυτό. Κύριε Μαριά, παρακαλώ. Την 683 και την 676 και μετά την 049. Κυρία Πρόεδρε, οι αναφορές αυτές ε, αναφέρονται στην ίδια την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Ε, αναφέρονται από μια σκοπιά που εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ από τη, στη σκοπιά που θέτουν οι, οι αναφέροντες. Ε, έχουν τη δικιά τους άποψη και βλέπουν τα ζητήματα. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε την άσκηση της νομισματικής πολιτικής διότι υπάρχουν και άλλες πλευρές, φερειπίν ε, οι πολίτες στην Ελλάδα ή στον Ευρωπαϊκό Νότο επίσης μπορεί να διαφωνούν με την άσκηση της νομισματικής πολιτικής από πλευράς Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως εδώ πρέπει να δούμε πρώτον ότι η, βεβαίως η άσκηση της νομισματικής πολιτικής είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ευρωσυστήματος όχι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών μέρος της οποίας είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό το ξεκαθαρίζω για να απαντήσω στην Κομισιόν. Διότι υπάρχει μια λάθος αντίληψη ότι η νομισματική πολιτική είναι μονοπόλιο του κυρίου Ντράγκη. Δεν είναι έτσι. Είναι μονοπόλιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών που είναι ένα σύστημα αποκεντρωμένο και δεν είναι σύστημα συγκεντροποιημένο. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση επειδή δεν είναι μια ε, τέλεια νομισματική περιοχή, είναι βέβαιο ότι θα έχει οικονομίες οι οποίες αναπτύσσονται, όπως εν προκειμένου η Γερμανία, η Ολλανδία, η Γαλλία κλπ. και οικονομίες οι οποίες μένουν πίσω. Είχα θέσει λοιπόν το θέμα αυτό στον κύριο Ντράγκη στο πλαίσιο του νομισματικού διαλόγου πριν από τρει μήνε, τέσσερι, αλλά εκεί δεν είχαμε το χρόνο να το συζητήσουμε. Διότι μπαίνει το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να εφαρμόσεις ένα ενιαίο κουστούμι μια νομισματικής πολιτικής για οικονομίες χωρών οι οποίες είναι σε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης και είναι επίσης και σε διαφορετική φάση. Δηλαδή σε φάση ανάπτυξης ε, η Γερμανία και σε φάση ε, όπου έχει πολλά προβλήματα με την ε, ανεργία, με τη φτώχεια η Ελλάδα ή η Ιταλία είχα κάνει την εξή πρόταση και κατά την έννοια αυτή έχει μια αξία η συζήτηση, γιατί θα πρέπει να πάμε σε μια αλλαγή και τη συνθήκη και τη Ευρωζώνη, ότι προφανώ η Κεντρική Τράπεζα και το Κεντρικό Σύστημα να μπορεί να εφαρμόσει μια ενιαία νομισματική πολιτική, η οποία να έχει εργαλεία, φερπίν σε μια φάση όπου η οικονομία της Ευρώπης αναπτύσσεται. Αλλά να επιτρέπεται σε χώρες οι οποίες βρίσκονται σε απόκληση από την οικονομική πολιτική σε χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, σε χώρες οι οποίες έχουν βγει μόλις τώρα από τα μνημόνια, να επιτρέπεται στις δικές τους εθνικές κεντρικές τράπεζες να ασκήσουν δική τους νομισματική πολιτική μέχρι του ύψους του ποσοστού που έχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα ο ισολογισμός της Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωσυστήματος είναι 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Φέρνω ένα παράδειγμα. Η Ελλάδα έχει μόνο 2% ε, μετοχικό κεφάλαιο. Να μπορεί η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος να ασκεί ανεξάρτητη νομισματική πολιτική στο ύψος του 2%. Δηλαδή σε επίπεδο 70 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και με αυτόν τον τρόπο να μην δεσμεύεται να ακολουθεί την κεντρική γραμμή η οποία λαμβάνει υπόψη και σωστά λαμβάνει υπόψη τις οικονομίες των αναπτυγμένων χωρών αλλά κάνοντας μια διαφορετική νομισματική πολιτική αυτές οι χώρες που είναι σε πρόβλημα και βγήκαν από τα μνημόνια να μπορούν φερπίν να ενισχύσουν την παραγωγή, να ενισχύσουν την ανάπτυξη, να ενισχύσουν τα θέματα της απασχόλησης ενώ η κεντρική πολιτική μπορεί να είναι διαφορετική. Άρα λοιπόν έχει αξία η αναφορά αυτή η οποία τίθεται υπόψη μας, διότι βάζει ένα θεμελιώδες ζήτημα. Μπορεί αυτή η Ευρωζώνη να προχωρήσει με αυτούς τους όρους που ξέρουμε. Μια Ευρωζώνη που στην ουσία κερδίζει μεγάλο μέρος κυρίως η ισχυρή οικονομία, δηλαδή κατά κύριο λόγο η Γερμανία, παρότι είναι Γερμανός ο αναφέρον και διαφωνεί. Μήπως πρέπει να αλλάξει η δομή. Μπορείς να έχεις μια Ευρωζώνη που βοηθά πλεονάσματα εμπορικά 8,9% στη Γερμανία, τα οποία δεν μοιράζει καν η Γερμανία στο γερμανικό λαό. Γι' αυτό και είδαμε τα αποτελέσματα τα τελευταία των εκλογών. Επομένως, κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον η αναφορά, όχι ως προς την πολιτική και την ουσία που θέτει, θέλει μια άλλη νομισματική πολιτική, αλλά στη δομή που πρέπει να έχει η νομισματική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως έχουμε και κάνει και ε, έχει ψηφίσει το κοινοβούλιο μας, νομίζω την τελευταία συνεδρίασε στο Στρασβούργο, για τα θέματα διαφάνειας. Όπου στα θέματα διαφάνειας, νομίζω ήταν η εισήγηση του κ. Γκίγκολτ, εκεί πραγματικά τίθενται ζητήματα για το πώ πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και στη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να μείνουν ανοιχτέ και να σταλούν στην Επιτροπή οικονομική και νομισματική πολιτική ω ένα στοιχείο διαλόγου, ανησυχία για το πώ πρέπει να οργανωθεί στο μέλλον η νομισματική πολιτική και για το πώ πρέπει να κάνουμε κάποιε αλλαγές προς την α ή τη β κατεύθυνση. Άρα είναι ένα στοιχείο, θα έλεγα, αναφορών γενικού προβληματισμού που δίνουν την ευκαιρία να συζητήσουμε σοβαρά θέματα και να αναπτύξει ο καθένας τις δικές του προτάσεις για το πώς μπορεί να προχωρήσει η Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. I think that what we just... Νομίζω ότι αυτό το οποίο μόλις αποφασίσαμε στην αναφορά 91 και 161 ε, περαιτέρω δράσεις, επιστολή κλπ. θα μπορούσε να επαρκεί. Και κατά την άποψή μου αυτή η αναφορά θα μπορούσε να κλείσει διότι η, τα θέματα της διαφάνειας απαντώνται στις προηγούμενες και νομίζω ότι κατ' ουσίαν και αυτή και οι επόμενες δύο αναφορές θα μπορούσαν να κλείσουν. Μπορείτε να αφήσετε ανοιχτή μόνο την 676 για τη μονομερή και αντιδημοκρατική νομισματική πολιτική. Αυτό είναι διαφορετικό. Μπορεί να μείνει open, να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Και η άλλη αναφορά που συγκεκριμενοποιεί το θέμα των επιτοκίων κλπ. ίσως θα μπορούσε να κλείσει όπως λέτε. Εντάξει, εντάξει. Okay, we do that. The, so the petition... Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Η 683 κατά την άποψή μου πρέπει να κλείσει, όπως επίσης και η 429 και μετά θα κρατήσουμε την 676, την 161 και την 91 μαζί και Η 429, 9, η τελευταία, είναι, πρέπει να μείνει ανοιχτή γιατί αφορά θέματα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτή είναι τελείως διαφορετική, δεν τη συζητήσαμε. Και νομίζω ότι αυτή πρέπει να μείνει ανοιχτή, διότι αφορά και δικαιώματα των καταναλωτών και δικαιώματα των πολιτών και επομένως κατά τη γνώμη μου είναι πολύ πιο σοβαρή αυτή η υπόθεση σε αυτή τη φάση. Πιστεύω λοιπόν ότι και αυτή πρέπει να μείνει ανοιχτή και την οποία δεν συζητήσαμε. Δεν άκουσα την άποψη της Κομισιόν σε αυτή. Στην 429 του 17 δεν μας είπε την άποψη της Κομισιόν. Ε, ακριβώς. Ακριβώς. Θα, θα ακούσουμε αυτό. I invite you. Σας ε, ζητώ λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια και για την 429 για να έχουμε και την εικόνα, την άποψή σας και γι' αυτό. Συγγνώμη, το παρέλειψα προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ. Για να συνοψίσω με δύο λόγια, ο αναφέρον ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναφέρει τη θέση της για την ε, ε, άμεση παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ε, λειτουργίας των πιστοτικών ιδρυμάτων και ο, για να αλλάξει το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα και θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από πλευρά Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά την εφαρμογή τη νομισματική πολιτική. Ο κύριο ε, Μαριά ε, θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική είναι αποκεντρωμένη. συγγνώμη που δεν το ανέφερα αυτό προηγουμένω. Επαναλαμβάνουμε αυτά που σας είπαμε και προηγουμένως. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ανεξάρτητη στην ε, νομισματική πολιτική και εμείς σεβόμαστε πλήρως την ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Θεωρούμε λοιπόν ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να το απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ. Ναι, και γι' αυτό ακριβώς και εγώ θεώρησα ότι θα μπορούσε να κλείσει το θέμα. Ε, αλλά ο κύριος Μαριάς ε, να μας πει την άποψή του. Η τελευταία αναφορά, έτσι όπως την βάζουν οι αναφέροντες, έχει σχέση και με τις τελευταίες ρυθμίσεις που θέλει να κάνει ο κύριος Ντράγκη έναντι των τραπεζών για, για τα θέματα των κόκκινων δανείων. Δηλαδή τις υποχρεώνει να εγγράψουν στον ισολογισμό τους, όπως είπα, κονδύλια για τη διασφάλιση των κόκκινων δανείων. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες Υπάρχει η επιστολή του κυρίου Ταγιάννη, επομένως ε, πρέπει κατά την άποψή μου η μόνη αναφορά που να κλείσει είναι η 683. Οι υπόλοιπε αναφορές να μείνουν ανοιχτέ και να ακολουθήσουμε την πρόταση που είπατε, να του στείλουμε επιστολή κτλ. Και, και το θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μάλλον ε, της, του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων από την Κεντρική Τράπεζα είναι στον πυρήνα το, και του προβληματισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτών. Επομένω, πρέπει να μείνει ανοιχτή. Άρα, η πρόταση, κυρία Πρόεδρε, είναι όπω είπατε στι αναφορέ όλε να επιστολεί προ την Κεντρική Τράπεζα κλπ. Και, την 683 πράγματι να την κλείσουμε όπω ε, προτείνατε. Ωραία. Κλείνουμε την 683, αλλά κρατάμε ανοιχτές τις υπόλοιπες και θα παραμείνουν ανοιχτές εν αναμονή και της ψηφοφορία στην Ολομέλεια που θα γίνει σε λίγες μέρες. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Ε, έχουμε πολλή δουλειά όμως τώρα γιατί ε, πρέπει να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για διάφορα θέματα. Όπως είπα προηγουμένως, ε, επομένως αυτό και θα κάνουμε και να κλείσουμε το θέμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτως ή άλλως έχουν κλείσει και οι τράπεζες τέτοια ώρα. Αν κλείσει η τράπεζα θα έχουμε πρόβλημα με το ευρώ. Λέει ο κύριος Μαριάς. Πάμε στο σημείο 20. Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Και ας προχωρήσουμε στην επόμενη γνωμοδότηση. Σας ευχαριστούμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας βοηθήσατε να διευκρινίσουμε αυτά τα δύσκολα ζητήματα. Θα επανέλθουμε. Ε, είμαι βέβαιη γι' αυτό. Γνωμοδότηση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωτών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2016. Η συγητής είναι ο κύριος Ρεμπέγκα. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ε, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, η γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο θεματολόγιο μας κάθε χρόνο. Ε, αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και όπως κάθε χρόνο και φέτος η ε, έκθεση αυτή θα είναι πολύ πλήρης και γεμάτη στοιχεία. Θεώρησα ότι η ΠΕΤΗ μπορεί να συμβάλλει, ε, να επιφέρει προστιθέμενη αξία στην ε, έκθεση αυτή, συμπεριλαμβάνοντας θέματα που σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναφέρθηκαν πιο συχνά στις αναφορές του το 2016. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω τα θέματα που θύχτηκαν πιο ε, συχνά. Από τις 1569 ε, αναφορέ, αναφορές, οι 254 ε, αναφέρονταν στα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα θέματα κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα από την ελεύθερη κινητικότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία και τα σχετικά δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντος, ελευθερία έκφρασης και ισότητα των φύλων. Καθότι όμως ε, ε, είχα περιορισμό όσον αφορά τον ε, αριθμό των λέξεων στη γνωμοδότηση, έπρεπε να κάνω μια επιλογή. Έχω συμπεριλάβει λοιπόν στη γνωμοδότησή μου τα εξή θέματα. Ως αποτέλεσμα του Brexit λάβαμε αρκετές αναφορές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο που φοβούνται μην απολέσουν την ευρωπαϊκή ηθαγένεια και ότι θα επηρεαστεί το δικαίωμα ελευθερίας τους. Ε, γνωρίζετε ότι αυτό είναι μια από τις προτεραιότητες της διαπραγματευτικής μας ομάδας ε, στο Brexit. Επίσης, σε μεγάλος αριθμός αφορούσε ε, τις συνθήκες κράτησης των των φυλακισμένων. Αυτό είναι θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών. Πιστεύω όμως ωστόσο ότι θα πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τις συνθήκες ε, κράτησης ε, και να διασφαλίσουν το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων για τους φυλακισμένους. Άλλο σημαντικό θέμα είναι ε, η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα ε, διασφάλιση των δικαιωμάτων τους ε, και δικαίωμα στην φροντίδα και το κράτος ε, θα πρέπει να λαμβάνει πρωτίστως υπόψη το ύψιστο συμφέρον του παιδιού και να φροντίσει να υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια στις πολιτικές στον τομέα αυτών. Επίσης είχαμε θέματα κοινωνικής ασφάλειας, πρόσβαση στη ιατρική περίθαλψη και σε φάρμακα. Η Επιτροπή μας ε, το 2016 οργάνωσε εργαστήρι για την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και φάρμακα και είναι ε, λυπηρό το ότι ε, πολλοί πολίτες μας δεν έχουν τέτοια πρόσβαση. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρξει σωστή συνεργασία όσον αφορά τις τιμές και την ανταλλαγή πληροφοριών στα θέματα αυτά. Επίσης, ε, τονίζω την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος ε, και την ανάγκη να υπάρχουν ολοκληρωμένες πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεδομένου ότι πολλές ε, αναφορές που λαμβάνουμε αναφέρονται ακριβώς στο θέμα αυτό. Συνολικά το 17% των αναφορών που έχουν να κάνουν με, το, με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επίσης, η ισότητα των δύο φύλων και ελευθερία έκφρασης. Δεν θα πρέπει να περιορίζονται αυτά τα δικαιώματα. Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι το θέμα της προστασίας ε, των καταναλωτών. Σύμφωνα με τον ε, χάρτη των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο πολλών αναφορών το 2016, ιδιαίτερα στον τομέα τον τραπεζικό που έχει να κάνει με τα δάνεια. Ε, κυρία Πρόεδρε, ελπίζω ότι η γνωμοδότησή μου αυτή θα συμβάλλει στη βελτίωση ε, της ε, ζωής των Ευρωπαίων πολιτών και να σας θυμίσω ότι η προθεσμία την κατάσταση τροπολογιών είναι η 16η Οκτωβρίου του 2017. Προσλέβω στην συνεργασία με τους συναδέρφους. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είναι παρόντε άλλοι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή. Ένα συνάδελφο έχει το λόγο. Θα θέλατε να... Ε, είναι παρόν. Ε, Μήπω θα θέλατε να πάρετε το λόγο. Όχι. Πρόεδρο, ε, άρα μόνο εγώ απομένω. Θα ήθελα να καλέσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Στόκολ, να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρεμπέκα για το σχέδιο γνωμοδότησή του. Όλα τα θέματα που αναφέρατε είναι ιδιαίτερα επίκαιρα. Ε, Δυστυχώ είναι αρκετά τα θέματα αυτά, αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και απομένουν πολλά να γίνουν όσον αφορά την προστασία των θεμελιωτών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το πρωί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ε, έκθεσή τη ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που είναι επί αρμόδια για την έκθεση αυτή. Ο εισηγητής ήταν παρόν και θα ήθελα να τονίσω ε, τα βασικά στοιχεία της παρέμβασης της Επιτροπής ε, σήμερα το πρωί. Καταρχάς ε, η Ένωσή μας βασίζεται σε αξίες και ο χάρτης είναι κατάλογος νομικών δεσμεύσεων, δεν είναι κατάλογος επιθυμιών. Ε, η δεύτερη παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ήταν ότι η εξωτερική αυτόνομη εποπτεία είναι πάρα πολύ σημαντική και στην έκθεση τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος των εθνικών δικαστηρίων και καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, ο ρόλος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των οργανισμών για την υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Και τρίτον, ε, το σχέδιο έκθεσης ε, ε, τονίζει ακριβώς το θέμα των κοινωνικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την διαδικασία. Επικεντρώνεται όμως και σε κάποιους τομείς στους οποίους θα πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες όπως είναι η ισότητα των δύο φύλων, η Ρωμά, η μετανάστευση, τα δικαιώματα των παιδιών. Και να σας ε, θυμίσω δύο εκδηλώσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και που σχετίζονται με τα θέματα που θίγεται στην γνωμοδότηση. Στις 6, 7 και 8 Νοεμβρίου έχουμε το Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού που θα επικεντρωθεί ε, στην κράτηση παιδιών και τις εναλλακτικές λύσεις και ε, την ε, τρίτη ε, συνάντηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που θα πραγματοποιηθεί επίσης τον Νοέμβριο που αυτή τη φορά επικεντρώνεται στα δικαιώματα των γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξαναρωτήσω τον κύριο Ρεμπέκα, υπάρχει κάτι που θέλετε να προσθέσετε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, για τις πληροφορίες αυτές. Θα ήθελα ταυτόχρονα να σας διαβεβαιώσω ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, πρέπει να ισχύουν για όλους και αγωνιζόμαστε ακριβώς γι' αυτό. Ακόμα και όταν ε, έχουμε διαφορές, διαφορετικές πολιτικές απόψεις, εδώ μιλάμε για κάτι που δεν είναι θέμα πολιτικών απόψεων, αξίζει πολύ περισσότερη προσοχή από την πλευρά μας και σας διαβεβαιώ ότι Είμαι ανοιχτός σε συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, να επαναλάβω ότι η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι στις 3 η ώρα, στις 16 Οκτωβρίου, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή. Και έτσι... Ολοκληρώνουμε τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Εύχομαι σε όλους καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.